Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές ε, φίλες και αγαπητοί φίλοι, έχουμε την ευκαιρία να πούμε αγαπητές ε, φίλες και αγαπητοί φίλοι. Χωρίς να το λέμε αυτό μόνο για το Θεαθήνε, μόνο επίσημα ή από ευγένεια γιατί ακριβώς επειδή είμαι πάρα πολύ καιρό αρμόδιος για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, βλέπω πολλά οικία πρόσωπα και πολύ σημαντικούς ε, συναδέρφους, αλλά πάνω απ' όλα πολύ καλούς φίλους και φίλες. τους οποίους ε, χαιρετίζω εγκάρδια και με ιδιαίτερη στοργή. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ευκαιρία που έχουμε να σας υποδεχτούμε εδώ όλες και όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνάντηση αυτή με θέμα το ρόλο των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Έχουμε την ε, ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη Τη διοργάνωση, ο αντιπρόεδρος Ότμαρ και ο υποφαινόμενο. γιατί είμαστε εμεί οι δύο αντιπρόεδροι που στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την ευθύνη ή μοιραζόμαστε την ευθύνη των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε μια αρκετά φορτωμένη μερίσια διάταξη που βρήθη πολύ σημαντικών θεμάτων και ο κύριος Κάρας στην ουσία θα αναφερθεί στην ουσία της σημερινής συνάντησης, γιατί εκείνος ανέλαβε όλες τις προετοιμασίες. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνω αυτή την σύντομη εισαγωγή, να σας απευθύνω χαιρετισμό και να κάνω και κάποια πιο γενικά σχόλια. Γιατί έχουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ ικανοποιητική η εκπροσώπηση εδώ. Πολλά εθνικά κοινοβούλια έστειλαν εκπροσώπους σε αυτή τη συνεδρίαση. Και μάλιστα έχουμε και συναδέλφους με υψηλά αξιώματα, όχι μόνο σε Προεδρία Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά και σε σημαντικές επιτροπές Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε λοιπόν και Προέδρους Επιτροπών. Και επίσης με ιδιαίτερη ικανοποίηση ε, θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό και σε πολλούς αξιωματούχους και υπαλλήλους ε, των κοινοβουλίων μας και μάλιστα με μερικούς από αυτούς έχουμε πολύ μακροχρόνια σχέση γιατί σε πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούμε ιδιαίτερα στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ η συνεργασία μας με τους υπαλλήλους αυτούς είναι πάντα πολύ στενή και πολύ χρήσιμη. Χαιρετίζω λοιπόν και τους ε, υπαλλήλους των κοινοβουλίων και τους ε, υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρόνια ολόκληρα μας ε, συνοδεύουν σε αυτές τις συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και επίσης να καλωσορίσω και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Εκπρόσωποι των διοικήσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων στην διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί μερικά κοινοβούλια έχουν δύο βουλές, δύο σώματα. Αλλά δεν είναι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων. Είναι, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων είναι μόνο βουλευτές. Οι υπόλοιποι είναι αξιωματούχοι, οι υπάλληλοι στα κοινοβούλια αυτά. Όπω είπα, ο φίλος Ότμαρ Κάρας ε, θα περάσει την ουσία της σημερινής συζήτησης. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω κάτι που ήδη γνωρίζετε, ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλοι, όλοι μας ανησυχούμε κάπως από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από διάφορες δημοσκοπήσεις και από το Ευρωβαρόμετρο πληροφορίες που μας φέρουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Δηλαδή με το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα σε αυτές τις ευρωεκλογέ θα έχουμε άνευ προηγουμένου αποχή. Και μάλιστα πολύ ανησυχητική αποχή. Ή, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, θα έχουμε τόσο ισχνή συμμετοχή που θα είναι πολύ ανησυχητική. Τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε δεν περιορίζουν αυτή την απώλεια στα κοινοτικά θεσμικά όργανα μόνο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα στοιχεία που μελετάμε δείχνουν μία αυξανόμενη απομάκρυνση των Ευρωπαίων πολιτών, μία αποσύνδεση, αποστασιοποίηση των Ευρωπαίων Ευρωπαίων πολιτών από τις εκλογές και από την ε, εκπροσώπησή τους στο κράτος δικαίου. Έχουμε δηλαδή μια αποστασιοποίηση των πολιτών ή όλο ε, μια αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς στη δημοκρατία και στην πολιτική γενικά. Αυτά δυστυχώς τα συμπεράσματα μας προβάλλουν τα στοιχεία που λαμβάνουμε και ακριβώς μας δημιουργούν μια τεράστια πρόκληση για όλους μας και ε, για μας που βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην συνεδρίαση αυτή. Και από αυτή την άποψη και λαμβάνοντας υπόψη αυτή την μεγάλη ανησυχία έχει μεγάλη σημασία αυτά που θα, έχουν μεγάλη σημασία αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα εδώ. Και θα ολοκληρώσω με ένα άλλο στοιχείο που με επηρεάζει και προσωπικά, γιατί εκτός από τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, και μάλιστα είναι, ε, έχω αναλάβει και ένα άλλο θέμα, ένα συναρπαστικό ζήτημα που είναι το η δημιουργία του οίκου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είμαι συναρμόδιος με το Hans Gerd Πέτερινγκ, που ήταν πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νυν πρόεδρος του Ιδρύματος Κόνερα Ταντενάουερ στη Γερμανία. Και αυτό πραγματικά, αυτό το καθήκον είναι το πιο συναρπαστικά. Αυτή η αρμοδιότητα για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πέραν όμως αυτής της αρμοδιότητας, έχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θέματα της πολυγλωσσίας, δηλαδή της μετάφρασης και της διερμηνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο στον κόσμο που από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε με 24 ε, γλώσσες, που είναι 24 επίσημες γλώσσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακριβώς επειδή είμαστε ή έχουμε την αξίωση να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο παίκτη. Εκτός από, τα εκτός από τις 24 αυτές επίσημες γλώσσες, χρησιμοποιούμε και γλώσσες και άλλων παγκοσμίων ε, ε, σημαντικών εταίρων και παικτών, με τους οποίους ε, συμμεριζόμαστε την παγκόσμια ευθύνη για την ειρήνη, για την κοινωνική πρόοδο και τόσα άλλα σημαντικά θέματα. Πολύ συχνά λοιπόν χρησιμοποιούμε τα ρωσικά, τα αραβικά, τα κινέζικα στις συνεδριάσεις που είναι γλώσσες των άλλων σημαντικών παικτών στο παγκόσμιο προσκήνιο. Επίσης και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ακούμε και να μιλάμε όλες τις γλώσσες των εκπροσώπων εδώ. Και υπάρχουν εδώ έντονες πιέσεις, γιατί μερικοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τα κονδύλια μας, να ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα και υπάρχουν πολύ ισχυρέ δυνάμεις που προσπαθούν πάση θυσία να μας περικόψουν τις δαπάνες. Εδώ όμως ο καθένας μιλάει τη γλώσσα του γιατί είναι σημαντικό και οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας να μπορούν να ακούν ό,τι διαμείβεται εδώ στην μητρική τους γλώσσα. Το θέμα δεν είναι να μιλάμε εμεί τη μητρική μα γλώσσα. Το θέμα είναι να ακούν στην γλώσσα του οι συμπολίτε μα, οι συμπατριώτε μα. Και αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή το θέμα τη εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, τη εμπιστοσύνη του στη δημοκρατία, το θέμα αυτό αναφυσβήτητα συνδέεται άρρηκτα με το, τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να παρακολουθούν στη μητρική τους γλώσσα τις συζητήσεις εδώ. Γιατί 80% των Ευρωπαίων πολιτών μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. Δεν γνωρίζουν καμία ξένη γλώσσα. Το 80% των συμπολιτών μας μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα. και οι Βρετανοί το ίδιο. Μόνο ότι η δική τους γλώσσα μιλάνε. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό λοιπόν, οπότε δεν είναι καμία πολυτέλεια, καμία κεντρικότητα και καμία φοβερή πρωτοτυπία όπως την παρουσιάζουν μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπερβάλλουν και στο κόστος, γιατί οι δαπάνες της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα ουσιαστικά στοιχίζει σε κάθε πολίτη ένα καφέ το χρόνο. Είναι περίπου 500, 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 500 εκατομμύρια είναι και κάτι και ουσιαστικά ένα ευρώ το χρόνο στοιχίζει τον κάθε πολίτη. Ένα καφέ ουσιαστικά η πολυγλωσία. Ενώ είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του και να ακούγεται στη γλώσσα του. Γιατί μιλούσαμε όλοι μία ή δύο γλώσσε μόνο που θα ήταν οι γλώσσε εργασία, δεν θα μπορούσαν να μα παρακολουθήσουν οι περισσότεροι συμπολίτε μα. Δεν θα δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι διαμείβεται εδώ και τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και θα ήθελα να χαιρετήσω και του διερμηνείς μα, που είναι σημαντικό εργαλείο στη δυνατότητα επικοινωνίας και στην δημοκρατική ταυτότητα του σχεδίου. Να χαιρετήσω και τους τεχνικούς που επίσης ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των πολύ περίπλοκων μηχανισμών. Μάλιστα έχουμε συμφωνίες με 140 πανεπιστήμια που διοργανώνουν σεμινάρια, μαθήματα επιμόρφωσης και κατάρτισης διερμηνέων. Είναι σημαντικό λοιπόν ο καθένας να μιλά τη γνώση που θέλει και έχοντας υπόψη ότι ό,τι λέμε μεταδίδεται απευθείας σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν από πλευράς μου και με μεγάλο ενδιαφέρον θα δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ότμαρ Κάρας, για να σας εξηγήσει τις προετοιμασίες αυτής της διάσκεψης και το τι προσδοκούμε από αυτήν. Ότμαρ, έχεις το λόγο. Αγαπητέ Μαρτίνες, ε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου και μένα να σας ε, καλωσορίσω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το Κοινοβούλιο των Πολιτών της Ευρώπης. υποκανονικές συνθήκες συναντιόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για θέματα όπου έχουμε και οι δύο πλευρές αρμοδιότητες. Δηλαδή πριν από λίγες μόνο εβδομάδες εδώ ακριβώς σε, αυτό το χώρο διοργανώσαμε την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα από την Ελληνική Προεδρία και εγκαινιάσαμε τις συζητήσεις σε δύο τομείς αφενός όσον αφορά το ε, Δημοσιονομικό Σύμφωνο και αφετέρου τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σε αυτές λοιπόν τις ε, συναντήσεις, πρέπει να σας πω, μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι δεν βρισκόμαστε ακόμα στο ίδιο σκάφος, διότι βρισκόμαστε περισσότερο σε μία φάση όπου είμαστε επιφυλακτικοί η μία πλευρά απέναντι στην άλλη φέρουμε όλοι μας ε, τις ευθύνες μας απέναντι στην κρίση και την παγκοσμιοποίηση και καλούμεθα να δώσουμε απάντηση. Στη σημερινή λοιπόν ε, συνδιάσκεψη σας καλέσαμε για να συζητήσουμε θέματα που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές και μια τέτοια κοινή υπόθεση που αφορά όλα τα κοινοβούλια μια τέτοια λοιπόν κοινή υπόθεση είναι η ενίσχυση των εθνικών κοινοβουλίων, η αντιμετώπιση των κοινοβουλίων ως ε, κοινοβούλια πολιτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενίσχυση των κοινοβουλίων στη σημερινή εποχή της ε, παγκοσμιοποίησης. Γιατί μόνο με την ενίσχυση αυτή θα μπορέσουμε να βρούμε τις ε, απαντήσεις σε ερωτήματα όπως είναι η κρίση, η παγκοσμιοποίηση, ο εκδημοκρατισμός. Γιατί η προϋπόθεση όλων αυτών είναι η κοινοβουλευτική διάσταση που θα παρισφρήσει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε λοιπόν μια κοινή υπόθεση και αυτή η κοινή υπόθεση είναι ο ρόλος των κοινοβουλίων ενίδη εκπροσώπησης ε, των πολιτών, η ενίσχυση των κοινοβουλίων στην σημερινή δημοκρατία. Καλούμεθα να ορίσουμε το ρόλο μας και καλούμεθα να είμαστε πραγματικοί εκπρόσωποι των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία ε, λήψης αποφάσεων. Ο δικός μας ο ρόλος προφανώς επικύλει ανάλογα με την κάθε χώρα και υπάρχουν πολλές ε, εξελίξεις ε, όπου βλέπουμε ότι δεν επικρατεί η κοινοβουλευτική διάσταση στις ε, διαδικασίες αλλά επικρατεί περισσότερο η κυβερνητική βούληση. Η σημερινή λοιπόν συνάντησή μας θα έχει ως στόχο να προωθήσει αυτήν την κοινή μας υπόθεση, αυτόν το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο καθένας από εμά σε αυτή την ε, σημερινή Ευρώπη και στο σημερινό κόσμο. Επίσης, επιθυμώ να προσθέσω ότι σήμερα είμαστε 96 ημέρες πριν από τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές. Βεβαίως και τίθεται το θέμα της προσέλευσης στις εκλογές. Και αυτό ανέκαθεν ήταν ένα θέμα που αφορούσε τα κοινοβούλια και στήριζε την κοινοβουλευτική διάσταση. Όμως πλέον στις ε, σφιγμομετρήσεις βιώνουμε καθημερινά και το επισήμανε αυτό ο συνάδελφος ε, κύριος Μαρτίνες ότι υπάρχει μία άμεση σχέση ανάμεσα στη γνώση των πολιτών για το ρόλο των κοινοβουλίων, μια σχέση ανάμεσα σε αυτή τη γνώση και αφετέρου στην επιρροή που μπορεί να ασκήσει ένα κοινοβούλιο. Ο πολίτης επιθυμεί να γνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει ένας βουλευτής σε ένα κοινοβούλιο, την επιρροή που μπορεί να ασκεί και από εκεί εξαρτάται και η προσέλευση στις εκλογές. Όσο λοιπόν περισσότερα στοιχεία γνωρίζει ο πολίτης για, το ρόλο μας, για τη συμμετοχή μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η προσέλευση των πολιτών. Και τόσο περισσότερο περιορίζονται οι διαμαρτυρίες και ο λαϊκισμός. Και αυτό λοιπόν είναι κοινή υπόθεση για όλους μας. Κυρίες και κύριοι, στη τελική ανάλυση στην Ευρώπη ε, δεν είμαστε μόνο εμείς το διακύβευμα και γι' αυτό το λόγο ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Άντερσα Τζόνσον είναι ο κεντρικός ομιλητής της ε, συνάντησής μας ο οποίος ήρθε ακριβώς γι' αυτό το λόγο σε μας για να μας μιλήσει για το ρόλο μας στην σημερινή παγκοσμιοποίηση και στο πλαίσιο των ε, πολυμερών και διεθνών οργανισμών. Τον καλέσαμε για να συζητήσουμε για τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα και για να μπορέσουμε ή δυνατόν να ανταλλάξουμε βέλτιστες ε, πρακτικές. Κατά τις ε, προηγούμενες δεκαετίες οι κυβερνήσεις μας δήλωσαν συμμετοχή και συνέστησαν μάλιστα μια μεγάλη σειρά ε, πολυδιεθνών οργανισμών. Οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί, πολλοί εξ αυτών, συνδέονται μεταξύ τους με γραμματείες, με μηχανισμούς. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι μικροί άτυποι οργανισμοί και σε πολλούς από αυτούς τους ε, οργανισμούς ε, οι κυβερνήσεις ε, λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, αποφάσεις όμως οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλούς από αυτούς τους μικρούς οργανισμούς λαμβάνονται αποφάσεις που προκαταλαμβάνουν τη λειτουργία τόσο των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αναφέρομαι στην ρύθμιση για την εποπτεία τραπεζών, ρυθμίσεις παρήματος χάρη για τα πνευματικά δικαιώματα ή και ρυθμίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές ε, για την παραγωγή προϊόντα. Οι διεθνείς αυτοί οι οργανισμοί επηρεάζουν πάρα πολλές πτυχές της ε, καθημερινής μας ζωής και της ε, καθημερινότητάς μας. Αυτοί λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί είναι απαραίτητοι, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν συμβάλει στο να έρθουν πιο κοντά οι χώρες μας. Αυτή η παγκόσμια η πολιτική, η παγκοσμιοποίηση αν θέλετε, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κυβερνήσεις και σε διπλωμάτες. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό αυτές τις διαδικασίες να τις ε, ε, να τους δώσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση, να εκδημοκρατήσουμε αυτές τις διαδικασίες, να συμμετέχουν σε αυτές τόσο τα εθνικά όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Διεθνής Κοινοβουλευτική Ένωση και αυτή να συμμετέχει. Γιατί οι βουλευτές, όπως είμαστε εμείς, οι ερετοί εκπρόσωποι των πολιτών, εμείς λοιπόν καλούμεθα σε αυτές τις διαδικασίες να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο. Και ναι, ε, κατά το πρόσφατο ε, παρελθόν ε, οι οργανισμοί πολύ εξ αυτών πράγματι προσέλαβαν αυτή την ε, κοινοβουλευτική διάσταση, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο για πάρα πολλούς εξ αυτών. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα κύριο Τζόνσον για τη δική του την προσωπική συμβολή στις επαφές ε, στις οποίες καλλιέργησε έτσι ώστε πράγματι οι βουλευτές να γνωριστούν καλύτερα και να μπορέσουν να επιτρέψουν αυτή την συνεργασία των ε, διεθνών οργανισμών. Δεν καλούμεθα να επανανακαλύψουμε τον τροχό. Το μόνο το οποίο καλούμεθα να κάνουμε είναι να έχουμε στενή συνεργασία με διάφορα κοινοβούλια και να ε, προσαρμόσουμε τα καθήκοντά μας. Θέλω εξάλλου να σας πω Όπως είπε και ο συνάδελφός μας ε, ε, κύριος ε, Μαρτίνες ότι θα υπάρξουν αρκετοί, όπως ο συνάδελφός μου που δεν θα συμμετέχει πλέον στο επόμενο κοινοβούλιο. Γι' αυτό καλό να τον ευχαριστήσουμε τώρα, τον κύριο Μαρτίνες, για τη συμμετοχή του στην ΚΟΖΑΚ και επίσης και στις δραστηριότητες του για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ε, όλοι όσοι εν πάση περιπτώσει δεν θα είσαστε στην επόμενη, στο επόμενο κοινοβούλιο να βρείτε τους ε, αντάξιούς σας ε, διαδόχους για να συνεχιστούν οι εργασίες. Εγώ λοιπόν τάσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ του εκδημοκρατισμού και της ενίσχυσης του ρόλου των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή τη διεθνή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί όλο και περισσότερο λαμβάνονται υπερεθνικές αποφάσεις από τον ε, ΙΕ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το G8, από το G20. Οι αποφάσεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο δεν θα πρέπει να λαμβάνονται και κλεισμένα των θυρών, αλλά οι αποφάσεις αυτές ε, να υποβάλλονται σε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο. Και θέλω να σας πω το εξής. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, εργάζομαι για την αξιολόγηση της Τρόικα στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει έρευνες και έχουμε διαπιστώσει ότι περισσότερη δημοκρατία είναι απαραίτητο να υπάρξει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα αιρετά κοινοβούλια εκπροσωπούν τους πολίτες, άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί εκείνοι που θα συμπεριλαμβάνουν περισσότερο τα κοινοβούλια στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η Τρόικα είναι μια ειδική περίπτωση και η Τρόικα δεν προέκυψε ε, μετά από ε, νομιμοποίηση με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, να υπάρχει διαφάνεια, την συνθέτουμε και τη συνδυάζουμε, τα προγράμματα της Τρόικα τα συνδυάζουμε με την κοινοβουλευτική διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω, εμείς θα μεριμνήσουμε μακροπρόθεσμα να παρισφρήσει στην Τρόικα αυτό το κοινοτικό στοιχείο. Δεν σημαίνει ότι επικρίνουμε την παρούσα κατάσταση, απλά θέλουμε να υπάρξει εξέλιξη έτσι ώστε την εμπειρία που αποκομίζουμε από την έλλειψη δημοκρατίας σε αυτό τον οργανισμό, αυτή την έλλειψη δημοκρατίας στο μέλλον να την εξαλείψουμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας ένα μακρύ δρόμο μέχρι να επιτύχουμε την πλήρη διαφάνεια, την απόδοση ευθυνών, την ανάληψη ευθυνών σε διαδικασίε της αποφάσεων. Ο στόχος της εργασίας μας σήμερα είναι να υπάρξει μια γενική συζήτηση για τον μεταβαλλόμενο ρόλο των κοινοβουλίων, να αξιολογήσουμε ε, την επιρροή που μπορούμε να ασκούμε έτσι ώστε στο μέλλον να είμαστε πραγματικά πιο δυνατοί. Πώς μπορούμε ε, να έρθουμε πιο κοντά Υπάρχουν 32 πολυμερείς συνελεύσεις όπου συνεργαζόμαστε και σε αυτές τις συνελεύσεις ε, είναι μέλη είτε τα Εθνικά Κοινοβούλια είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να εισακούεται περισσότερο η φωνή μας και για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε την παγκοσμιοποίηση σε εσωτερικές εθνικές συζητήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να καθοδηγούμε και εμείς την παγκόσμια πολιτική. Με αυτή λοιπόν την έννοια ξεκινάει η συζήτηση, είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της συζήτησης σήμερα για να αναζητήσουμε μηχανισμούς ε, της ε, συνεργασίας. Γνωρίζετε λοιπόν ότι σήμερα μέχρι τις 12.30 μετά τη συζήτηση του Γενικού Γραμματέα θα συζητήσουμε. Το μεσημέρι προβλέπεται γεύμα για όλους μας και σε αυτό το μεσημεριανό γεύμα θα έχουμε τον κύριο Έλμαρ Μπροκ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας και είναι μέλος ε, των συνελεύσεων για το Σύνταγμα και για την, τον θεμελιώδη χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το απόγευμα θα συναντηθούμε από 14 μέχρι 15 και 40 για να δούμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διεθνή φόρουμ. Ε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και από τις 15 ε, και 40 μέχρι 15 και 20 είναι η δεύτερη συνεδρία που αφορά τις παγκόσμιες ε, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Αυτή τη συνεδρία, αυτής μάλλον, θα προεδρεύσει ο συνάδελφός μου κύριος Μαρτίνες. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να καλέσω τον κεντρικό μας ομιλητή, τον κύριο Τζόνσον, το Γενικό Γραμματέα της IPU, ο οποίος κυρίως Τζόνσον ε, έχει αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην ε, διεθνή διπλωματία, όπου και αν πάει κανείς στον κόσμο, παρίσταται πάντα ο ίδιος ε, και ανεξάρτητα με το που γίνονται συνέδρες, ο ίδιος είναι εκεί. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια. Εργάστηκε πάνω από 15 χρόνια στην ύπατη αρμοστία ε, προσφύγων. Μετά μπήκε το 1991 ε, στη γραμματεία της IPU και ο στόχος του είναι να εξελίξει την ε, IPU, να την ενισχύσει, να την εκδημοκρατήσει. Το 1998 εξελέγει Γενικός Γραμματέας ε, της IPU και έκτοτε έχει επανεκλεγεί τρεις φορές και φέτος την Άνοιξη θα παρετηθεί, δεν θα πάψει όμως να ενδιαφέρεται για την υπόθεση της ε, IPU. Έχει λοιπόν επιδείξει μια πολύ σημαντική σταδιοδρομία στον τομέα των διεθνών σχέσεων και της ε, κοινοβουλευτικής συνεργασίας και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Τζόνσον θα προσφέρει πολλά και ενδιαφέροντα κίνητρα για τη συζήτησή μας. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Σας δίνω το λόγο κύριε Τζόνσον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καράς Um, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ επίσης και τον Μιγγελ Άγχελ Μαρτίνες για τα επίσης καλά του λόγια. Παρασύρθηκα λίγο όταν πήρα την πρόσκληση και άρχισα να γράφω την ομιλία μου και έγραψα μια πολύ μεγάλη ομιλία. Ένα δοκίμιο θα έλεγε κανείς που ασχολείται και με τα θέματα τα εθνικά και με τα θέματα τα ευρωπαϊκά. Μπορείτε να τα διαβάσετε αν θέλετε, εγώ δεν θα το διαβάσω πάντως. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το ρόλο του κοινοβουλευτικού συστήματος στον παγκοσμιοποιημένο σήμερα κόσμο. Είναι οι κατάλληλες μορφές ε, αυτές εκπροσώπησης που έχουμε ε, σωστές η ανάπτυξη της δημοκρατίας παρακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την παγκοσμιοποίηση, έτσι ώστε για να καταλάβετε από πού προέρχομαι. Είναι αξιωματικό θα έλεγε κανείς ότι η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει πάρα πολλές αλλαγές στο σημερινό κόσμο. Δεν υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στα εσωτερικές υποθέσεις και τις εξωτερικές υποθέσεις. Τα περισσότερα από τα εσωτερικά θέματα μας απασχολούν όλους οι χώρες όλο και περισσότερο συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα. Το να δρά κανεί μόνος του γνωρίζεται πολύ καλά ότι δεν αποδίδει και σε τις άλλες και σε πάρα πολλούς τομείς στην Ευρώπη κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Για διάφορους λόγους, για διάφορους λόγους σε περιοχές όπως ε, η Ευρώπη τα κράτη άνοιξαν τις αγορές τους, τις οικονομίες τους αυτό σημαίνει ότι εκχώρησαν, έστω και επιμέρους, ένα τμήμα της κυριαρχίας τους σε μια κοινή περιφερειακή δομή. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από τη συνεργασία η οποία μπορεί να συμβεί σε επίπεδο παγκόσμιο ανάμεσα στα κράτη. Τα κράτη δεν έχουν αποφασίσει να μεταφέρουν κάποιες από τις εξουσίες τους και όλες συμμετέχουν κανονικά ισότιμα στις διεθνείς οργανώσεις που έχουν δημιουργήσει. Οι οργανώσεις αυτές είναι κυρίως διεθνή ε, διαπραγματευτικά φόρουμ αν και εξελίσσονται και ορισμένα προγράμματα στο εσωτερικό των κρατών. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά ακόμα πιο θολά τα σύνορα ανάμεσα στην εσωτερική πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, τα κυρίαρχα κράτη παραμένουν ο πυρήνας της διεθνούς τάξης και οι εξωτερικές υποθέσεις θεωρητικά τουλάχιστον παραμένουν αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας κάθε κράτους μέλους. Πέρα από αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την εξέλιξη των διακοινοβουλευτικών δομών. Η οργάνωση την οποία εγώ εκπροσωπώ, η Διακοινοβουλευτική Ένωση, δημιουργήθηκε εδώ και 125 χρόνια είναι η πρώτη αν θέλετε και η παλαιότερη φυσικά πολιτική οργάνωση στον κόσμο σε διεθνές επίπεδο. Η IPU λοιπόν ήταν το πρώτο παράδειγμα της πολυμερού συνεργασίας. Ιδρύθηκε στην βασική ιδέα ότι όταν υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε κράτη-μέλη ή και στο εσωτερικό τα πρέπει να βρίσκονται λύσεις με τον πολιτικό διάλογο. Η λέξη δημοκρατία δεν ήταν τμήμα του λεξιλογίου της IPU εκείνη την εποχή και στις πρώτες συνεδριάσεις της δεν θα την ακούσετε. Θα μπορούσε όμως να ακουστεί. Δεν την ονοματίζαμε τη δημοκρατία, αλλά παρόλα αυτά η οργάνωση υπεράσπιζε την ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει δημοκρατία και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Εκείνες τις παλιές εποχές υπήρχαν πολύ λίγες κοινοβουλευτικές οργανώσεις. Η σκανδιναβική, σκανδιναβική κοινοβουλευτική οργάνωση δημιουργήθηκε το 1907 και η κοινοβουλευτική οργάνωση της κοινοπολιτείας δημιουργήθηκε το 1911. Ήταν πολιτικές οργανώσεις, στήριζαν την ειρήνη, την πολιτική συνεργασία και δεν ήταν ούτε υπέθεταν ότι ήταν διεθνή τα κοινοβουλευτικά σώματα. <clears throat> Παρέμειναν τα πράγματα αυτά μέχρι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε είδαμε να εξελίσσονται τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Είδαμε νέες κοινοβουλευτικές συνελεύσεις να δημιουργούνται. Πολλές από αυτές συνόδευαν την δημιουργία περιφερειακών διακυβερνητικών μορφών οργάνωσης. Ε, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα καλό παράδειγμα. Δημιουργήθηκε το 1949 και ήταν μία από τις πρώτες κοινοβουλευτικές οντότητες διεθνούς συνεργασίας. Άλλες τέτοιες συνελεύσεις ε, παρέμειναν κάπως χαλαρές στη δομή τους με άλλες ε, οργανώσεις και απλά έδιναν την δυνατότητα συνεργασίας κοινοβουλευτικών από διάφορες χώρες σε συγκεκριμένους τομείς, σε συγκεκριμένες περιοχές. Στην ουσία ήταν κάτι ανάμεσα σε μη κυβερνητική οργάνωση και διακοινοβουλευτική οργάνωση. Βέβαια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου γύρω στο 90 υπήρχαν γύρω στις 50 οργανώσεις επίσημες ή ανεπίσημες διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Κάθε περιοχή είχε τις δικές της αυτόνομες ε, κοινοβουλευτικές οργανώσεις. 25 χρόνια μετά που βρισκόμαστε έχουν διπλασιαστεί οι αριθμοί. Ο πιο πρόσφατος κατάλογος που φτιάξαμε τον Ιανουάριο περιλαμβάνει 125 διακοινοβουλευτικές διεθνείς δομές και δεν είναι και πλήρης ο κατάλογος αυτός νομίζω. Μισές από αυτές, 54 από αυτές συνεργάζονται με δια, διακυβερνητικές μορφές συνεργασίας. 22 από αυτές το κάνουν αυτό επίσημα, εξαρτώνται επίσημα. Και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Αλλά κάθε περιοχή έχει τη δική της διακοινοβουλευτική δομή, χωρίς βέβαια να έχει τις αρμοδιότητες που έχετε εσείς σαν παράδειγμα. Πολλά τέτοια κοινοβουλευτικά σώματα περιλαμβάνονται στις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης. Οι υπόλοιπε είναι κάπως πιο χαλαρά συνδεδεμένες με τις διακυβερνητικές δομές. Συνεργάζονται παράλληλα με τη διακυβερνητική δομή, αλλά δεν έχουν υποχρεωτικά μια επίσημη σχέση με αυτήν που τους επιτρέπει να επηρεάζουν τη διακυβερνητική δομή. Σαν παράδειγμα η διακοινοβουλευτική συνέλευση του Συμφώνου Συνεργασίας ε, της ΑΠΟ Ανατολής μετά μιλάμε για τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά δίκτυα, τα NGO. Τα ασχολούνται με ό,τι θέμα μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν δίκτυα για την ανάπτυξη, για τον πληθυσμό, για το περιβάλλον, για την υγεία, για την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, την οικονομία, το εμπόριο, τον αφοπλισμό, ε, την καταπολέμηση των διακρίσεων κτλ. Και υπάρχει επίσης και μια ομάδα 30 τέτοιων οργανώσεων που ονομάζουμε αυτόνομες διακοινοβουλευτικές οργανώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν περιφερειακές δομές όπως το Ασιατικό Κοινοβούλιο, η Αραβική Διακοινοβουλευτική Ένωση, η διάσκεψη των προέδρων του της ομάδας των 8 και φυσικά και η δική μας IPU. Αυτές οι εξελίξεις αυτό το οποίο δείχνουν είναι ότι υπάρχει μια πραγματική ανάγκη ε, και συνεχίζεται να αυξάνεται αυτή η ανάγκη να ε, αναπαραχθεί σε διεθνές επίπεδο η οργάνωση των δομών και των εξουσιών σε εθνικό επίπεδο. Έχει νόημα κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ναι, όταν πράγματι βέβαια τα κράτη ε, εκχωρήσουν κάποιες από τις αρμοδιότητές τους στο διακυβερνητικό επίπεδο. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τις εθνικές κυβερνήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν παράδειγμα δείχνει ένα τέτοιο παράδειγμα και καθιστά την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαραίτητη είναι μια πραγματική διαδικασία ολοκλήρωσης. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ε, τότε θα πρέπει ίσως να δώσουμε μια διαφορετική απάντηση στο ερώτημα. Όσο λειτουργούν οι πολυμερείς οργανώσεις σαν φόρουμ διαπραγμάτευσης και αναφέρομαι εδώ στο ε, ΜΠΟΕ ή στα Ηνωμένα Έθνη, τότε απαιτείται δράση πάντα από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τα μέσα για την διασφάλιση της λογοδοσίας. Το θέμα είναι να ενσωματώσουν τη διάσταση αυτή στην καθημερινή τους εργασία. Η δημιουργία διεθνικών διακοινοβουλευτικών σωμάτων δεν έχει μεγάλο νόημα όταν δεν υπάρχει διεθνές εκτελεστικό σώμα το οποίο να ελέγχουν. Ένα, μια τέτοια βουλή, ένα τέτοιο κοινοβούλιο δεν θα έχει πραγματικές αρμοδιότητες και θα υπονομεύσει τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων. Θα κοστίσει πάρα πολύ χρήμα, κάτι το οποίο θα βλάψει τα υπόλοιπα κοινοβούλια και δεν θα είναι σε θέση να τηρήσει τις υποσχέσεις του και θα δώσει μια πολύ κακή εικόνα σύνεπως για τα κοινοβούλια γενικά και για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στο κοινό. Όταν εσείς ε, κύριε Μαρτίνες ήσασταν πρόεδρος της IPU ξεκινήσατε για πρώτη φορά στην ιστορία μια παγκόσμια συνάντηση προέδρων των κοινοβουλίων. Ε, συνεκλήθη στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι 150 πρόεδροι κοινοβουλίων που πήραν μέρος εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση και συζήτησαν το συγκεκριμένο θέμα. Για τους Προέδρους οι διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι αρμοδιότητα του εκτελεστικού σώματος, παρόλα αυτά μπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από τα κοινοβούλια. Με διαβούλευση και συνένεση των κοινοβουλίων πρέπει να υπάρχει επίσης και κοινοβουλευτική επικύρωση των συμφωνιών μέσω και εθνικών πολιτικών που συζητούνται στις, ε, στα κοινοβούλια και μέσω νόμων που χρηματοδοτούνται και ψηφίζονται από τα κοινοβούλια. Ώσπου να φτάσουμε στην εποχή όπου τα κράτη <coughs> θα εκχωρήσουν αρμοδιότητες στις διεθνείς διακοινοβουλευτικές ε, δομές, ε, τα περιθώρια δεν είναι πάρα πολλά. Η συνεργασία θα πρέπει να ξεκινήσει από τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Η τελευταία συνάντηση των Προέδρων το 2010 επιβεβαίωσε την τάση αυτή λέγοντας πως η εμπλοκή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διεθνή συνεργασία θα πρέπει να καθορίζει την καθημερινότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είπαν επίσης ότι η IPU είναι η καλύτερη διεθνής οργάνωση, η πιο κατάλληλη μάλλον, για την ε, εμπέδωση των σχέσεων ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς ξεκινάμε τώρα τις προετοιμασίες για την διάσκεψη των Προέδρων του 2015. Μια ομάδα Προέδρων, η οποία λειτουργεί σαν προπαρασκευαστική επιτροπή, συναντήθηκε τον Ιανουάριο. Οι απόψεις τους δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει. <coughs> Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζετε τη συζήτηση αυτή, την αντιμετωπίσατε το 2002 και 2003, όταν συζητήσατε τον καλύτερο τρόπο για μεγαλύτερη δημοκρατία στις εργασίες ε, του ΠΟΕ. Μετά από πολλές συναντήσεις και συζητήσεις καταλήξατε στο ότι ο πιο πρακτικός και πιο ευαίσθητος τρόπος αντιμετώπισης του θέματος είναι η δημιουργία μιας διακοινοβουλευτικής διαδικασίας η οποία να εδράζεται στα, εθνικά κοινοβούλια. Στόχος είναι η παρακολούθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων του ΠΟΕ διάλογος συνεχής με τους διαπραγματευτές, <coughs> ανταλλαγή εμπειριών και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών στα θέματα του διεθνούς εμπορίου και προσπάθεια επηρεασμού της κατεύθυνσης των συζητήσεων στον ΠΟΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η IPU είναι οι συνδιοργανωτές της ε, κοινοβουλευτικής διάσκεψης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου ε, και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το διάβημα αυτό και σήμερα συνεδριάζουμε στα γραφεία του ΠΟΕ. Έχουμε ε, ακροάσεις με το Διευθυντή του ΠΟΕ και με διαπραγματευτές από τις ε, κυβερνήσεις και έχουμε γίνει μια πολύ σεβαστή φωνή στη συζήτηση. Ε, συνεχίζουμε επίση και την προσέγγιση μα προ τα Ηνωμένα Έθνη και μάλιστα στην πρώτη διάσκεψη των ε, Προέδρων υλοποιήσαμε πολλά πράγματα. Καταρχήν είχαμε συμφωνία σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να διασφαλίσουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών ε, και των Εθνικών Κοινοβουλίων και κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται μέσω τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, τη IPU. Και αν δείτε το πρόσφατο ψήφισμα τη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων του Μαΐου του 2012 θα δείτε την τεράστια καμπή και την τεράστια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη σχέση αυτή. Σήμερα και τα κοινοβούλια έχουν έδρα έχουν μία θέση στο τραπέζι. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα νέα σώματα των Ηνωμένων Εθνών που δημιουργήθηκαν από το 2000 και μετά και έχετε και άμεση πρόσβαση σε αυτά και μπορείτε να συμμετέχετε σε όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε αυτή η σχέση να μεταφερθεί και σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχει άμεση επαφή και σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα σας και του δικού σας Εθνικού Κοινοβουλίου. Αυτή η σχέση είναι θεμελιώδου σημασία για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα πρέπει να κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια κτήμα τους ε, τα προγράμματα του ΟΗΕ και τις δραστηριότητες του ΟΗΕ. Αυτό μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο σημαντικό στις υπόλοιπε περιοχές του κόσμου εκ των πρώτη όψεω, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει αυτή η εθνική ιδιοκτησία, αυτό τα εθνικά κοινοβούλια να κάνουν κτήμα τους σε αυτά τα προγράμματα. Αλλιώς ε, οι συμφωνίες του ΟΗΕ δεν θα έχουν ε, πρακτική εφαρμογή και αποτέλεσμα αν δεν συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις και να ενημερώνονται. Πολλά προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και να είναι και τιμά του προπολογισμού, ώστε να εξασφαλίσει το, συμβούλιο, το Κοινοβούλιο συγγνώμη, διαφάνεια και λογοδοσία. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί μπορεί ο ΙΕ να είναι περισσότερο παρόν σε τέτοιε χώρες, αλλά ισχύει και για τις ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές κανονικά θα πρέπει να καταλήξουν σε συνολική συμφωνία, παγκόσμια συμφωνία το 2015. Αν στεθούμε επιτυχία, η συμφωνία αυτή θα αποφέρει τεράστιους καρπούς ε, για όλες τις χώρες. Θα έχουν όμως και σημαντικό τίμημα κάτι τέτοιε συμφωνίες. Είστε διατεθειμένοι να υπογράψετε μία λευκό επιταγή. Τα εθνικά κοινοβούλια, κατά τη γνώμη μας, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός μεταλλασσόμενου εθνικού διεθνού συστήματος που εξασφαλίζει δημοκρατική συμμετοχή, διαφάνεια και λογοδοσία σε πολλούς ε, διεθνείς οργανισμούς. Έχουμε σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Κατά τη γνώμη μου, η βασική πρόκληση για να λειτουργήσει το σύστημα αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Πώς θα οργανώσετε καλύτερα το έργο σας προκειμένου να διαδραματίσετε αποτελεσματικά το ρόλο σας. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό και σας ε, Παρακαλώ εδώ να εξετάσετε το πώς συμμετέχετε εσείς σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και προγράμματα. Θέλετε πραγματικά να διαδραματίσετε κάποιο ρόλο. Έχετε τέτοια αξίωση. Και αν ναι, πώς αντιμετωπίσετε το πρόβλημα το ότι οι διεθνείς σχέσεις και συμφωνίες δεν περιορίζονται πια στα παραδοσιακά, στις παραδοσιακές εξωτερικές υποθέσεις και λαμβάνουν χώρες, αφορούν κάθε σφαίρα της των, της ανθρώπινης προσπάθειας. Θα πρέπει λοιπόν να γεφυρωθεί αυτό το, το χάσμα μεταξύ του προγράμματος του Εθνικού Κοινοβουλίου και των λεγόμενων ε, εξωτερικών υποθέσεων. Πώς θα περιλάβετε στις καθημερινές σας εργασίες και αυτό το θέμα των εξωτερικών υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου αυτό το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά όλες τις χώρες του κόσμου για να σας ε, αναλύσω το διακύβευμα. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της αηφόρου ανάπτυξης μετά το 2015 και αν το γνωρίζετε πόσες εθνικές ε, βουλές ασχολούνται με το θέμα αυτό, πόσες ε, εθνικές ε, βουλές σχολιάζουν αυτά τα θέματα και παρέχουν πληροφορίες ή feedback στις διαπραγματεύσεις. Πώς θα εφαρμοστεί αυτή, αυτό το νέο πρόγραμμα, το νέο θεματολόγιο στις χώρες και στη δικιά σας φυσικά. Γνωρίζετε ότι υιοθετήθηκε μία δέσμη αναπτυξιακών στόχων το 2000 από τις διάφορες χώρες. Έχουμε ε, 7 στόχους για τις αναπτυσσόμενες χώρες και, μία, και ένα στόχο για τις αναπτυγμένες χώρες για να παρέχουν τους πόρους. Οι αναπτυξιακοί ε, στόχοι της χιλιετίας είναι σημαντικό τμήμα των διεθνών αναπτυξιακών προσπαθειών. Αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι θα ολοκληρωθούν το 2015 θα υιοθετηθεί ένα, μια νέα δέσμη αηφόρων αναπτυξιακών στόχων που θα λάβουν τη σκητάλη από τους προηγούμενους και όλες οι χώρες θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτούς τους ε, αναπτυξιακούς στόχους για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Και τον τελευταίο χρόνο, από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη, παρακινήσαμε τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να δείξουν ζωηρό ενδιαφέρον και να συζητήσουν αυτά τα θέματα στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να φροντίσουν να επηρεάσουν την όλη διαδικασία. Και μάλιστα γνωρίζω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Σχετική Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει συμπεριλάβει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εσείς, οι αδυναμίες ε, στην εφαρμογή των ε, αναπτυξιακών στόχων της ε, χιλιετίας αφορούν, σε αφορούν την έλλειψη εκπροσώπησης συμμετοχής και διαφάνειας. Σε καμία περίπτωση όμως ε, δεν ε, θα πρέπει κάτι τέτοιο να συνεχιστεί. Πιστεύω θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και εποπτεία. Γιατί αυτές οι αρχές βρίσκονται στην καρδιά αυτό που αποκαλούμε δημοκρατική διακυβέρνηση, που είναι η σύζευξη μεταξύ των δημοκρατικών αρχών με μια υγιή και αποτελεσματική διαδικασία λήψη αποφάσεων και εφαρμογή. Και υπό αυτό το πρίσμα, οι δημοκρατικέ αρχέ, αξίε και τα θεσμικά όργανα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να χαρακτηρίζουν και το αναπτυξιακό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί μετά το 2015. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί στο νέο αυτό πλαίσιο μετά το 2015 να μιλούμε μόνο για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Και μάλιστα το πλαίσιο των νέων αναπτυξιακών στόχων θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες και στα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί θα περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένους στόχους και δείκτες για την καταμέτρηση της πρόοδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων, θα δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και μεγαλύτερη στόχευση, θα συνοδεύεται από συγκέντρωση δεδομένων και έτσι θα επιτρέψει τα κοινοβούλια σα να ελέγξουν καλύτερα το κατά πόσο υλοποιούνται αυτοί οι στόχοι. Για όλου αυτού του λόγου έχει νόημα το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο να έχει και ένα στόχο που θα αφορά τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Έναν συνολικό στόχο που θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα περιορίζεται στις ικανότητες και στις λειτουργίες των κοινοβουλίων. Θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα περιλαμβάνεται και ένας τέτοιος στόχος. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σχέση με το το, το, το συλλογισμό της συμπερίληψη ενός στόχου δημοκρατικής διακυβέρνησης περισσότερο έχει σχέση με το γεγονός ότι οι κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή πραγματικότητα, χρειάζονται δηλαδή περισσότερη δημοκρατία στις διεθνείς σχέσεις και κάτι τέτοιο σημαίνει αναπόφευκτα μεγαλύτερη ανάμειξη των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν κατακλείδη λοιπόν θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες προκειμένου να βελτιωθεί η πολιτική εκπροσώπηση στις χώρες μας. Πιστεύω πάντως ότι σε διεθνές επίπεδο έχουμε ένα μοντέλο εργασίας για πολιτική εκπροσώπηση ώστε να λάβουμε καλύτερα υπόψη και να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Από πολλούς τρόπους, ε, από πολλές απόψεις είναι ε, ευρωπαϊκές οι ρίζες αυτού του μοντέλου. Και ενώ μερικές χώρες διαφυσβητούν τα θέματα τα εκτελεστικά, ε, κανονικά καθημερινά συζητάτε και δίνετε διαπραγματευτικές εντολές στους υπουργούς σας όταν εξετάζετε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και σας παροτρύνω αυτό το παράδειγμα να το μεταφέρετε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης θα πρότεινα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φανεί περισσότερο ρόλο σας και στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και ελπίζω ότι με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχιστεί το έργο του παλιού Κοινοβουλίου στη Διακοινοβουλευτική Ένωση αλλά δεν θα ήθελα να χάσετε μια ευκαιρία. Πιστεύω ότι μια πιο ενεργό συμμετοχή στη Διακοινοβουλευτική Ένωση ήταν επωφελής για όλους. Πιστεύω ότι έχετε το δυναμικό για να μπορέσει η δημοκρατία να παρακολουθεί την παγκοσμιοποίηση. Γιατί δεν χρειάζονται να δημιουργηθούν νέα θεσμικά όργανα. Ε, κατά τη γνώμη μου θα ήταν αναποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει τα δικά σας κοινοβούλια, που είναι αυτά που κατέχουν την εξουσία, να προσαρμοστούν και να διαδραματίσουν πολύ πιο ενεργό ρόλο σε θέματα διεθνούς συνεργασίας. Οπότε για να δημιουργηθεί το βιώσιμο αναπτυξιακό πλαίσιο και θεματολόγιο μετά το 2015 θα πρέπει ε, να αναλάβετε πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αυτή θα είναι πραγματικά η λιδία λίθος για όλα τα κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζόνσον. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτησή μας τώρα και πρώτος ε, ο μιλητής είναι από τον κύριο Σέντζο Σόζα Πίντο από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ και να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους φίλους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ε, χαιρετήσω και τον πρόεδρο Κάρας που πρόσφατα ήταν στην ε, Πορτογαλία, να το συγχαρώ για την έκθεσή του για το έργο της Τρόικα και διαπιστώσατε ότι δυστυχώς το έργο της Τρόικα διέφυγε οποιοδήποτε δημοκρατικού ελέγχου και από την πείρα που έχετε από το, την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου της Τρόικα στην Πορτογαλία ε, έχετε και κάποια εντύπωση για το πόσο δύσκολο είναι για τα, ευρωπαϊκά, για τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγξουν την παγκόσμια διαδικασία λήψη αποφάσεων. Η Πορτογαλία, όπως και άλλες χώρες μέλη, προσυπόγραψαν το ευρωπαϊκό σχέδιο και συμμετέχει σε βασικές ε, ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως είναι το ενιαίο νόμισμα. Γιατί πιστεύουμε ότι κάποιες ε, πτυχές ε, της εθνικής κυριαρχίας έπρεπε να εκχωρηθούν και χρειαζόμαστε μια υπερεθνική κυριαρχία, μια πανευρωπαϊκή κυριαρχία ώστε έτσι να διατηρηθούν ε, κάποιες πολιτικές, ε, να διασφαλιστεί η δημοκρατία και να παραμείνει αυτή στα χέρια των λαών. Και το ενίο νόμισμα ήταν ε, ένα εργαλείο που εξυπηρετούσε αυτό τον μεγαλοπρεπή και το μακρόπνο στόχο του ευρωπαϊκού σχεδίου, ώστε η δημοκρατία να ξεπεράσει τις απλές ε, αρχές της φιλελευθερωποίησης και της παγκοσμιοποίησης και να ξεπεράσει την ισχύ των παγκόσμιων αγορών ή των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η πορτογαλική εμπειρία των τελευταίων χρόνων δυστυχώς έδειξε την αποτυχία αυτού του στόχου. Η Πορτογαλία, όπως και άλλες χώρες, υπόκειται στη μόνη ουσιαστική κυριαρχία, που είναι η κυριαρχία δυστυχώς των τελευταιων χρονων δυστυχω εδειξε την αποτυχια αυτου του στοχου η πορτογαλια οπως και αλλες χωρες υποκειται στη μονη ουσιαστικη κυριαρχια που ειναι η κυριαρχια δυστυχω των αγορων Και στην ε, δημιουργία της πολιτικής για το ενιαίο νόμισμα χάσαμε τις εθνικές μας, τις κεντρικές μας τράπεζες, χάσαμε τη δυνατότητα να, ε, εκδίδουμε εμείς νόμισμα, ε, χάσαμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές και χάνουμε και τους ελάχιστους ε, απαραίτητους μηχανισμούς προάσπισης των ζωτικών μας συμφερόντων στα πλαίσια της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Και η παγκόσμια αντίδραση, η ευρωπαϊκή αντίδραση, η πολιτική αντίδραση, η μια δημοκρατική αντίδραση στην κρίση, μια αντίδραση και απάντηση δημοκρατικού ελέγχου δυστυχώς δεν υπάρχει. Οπότε δυστυχώς ο απολογισμός είναι αρνητικός. Και όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Πορτογαλία η πολιτική ζει για να ανακτήσει την μυθική εμπιστοσύνη των αγορών και ο μοναδικός στόχος που πριτανεύει, που εξαρτά και που επηρεάζει τις, πολιτικές που, τις επιλογές που γίνονται σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο ε, έχει δυστυχώς ολέθρια κοινωνικά αποτελέσματα και όχι μόνο κοινωνικά αποτελέσματα, γιατί εκεί έχουμε σημαντική παλιδρόμηση αλλά δυστυχώ και σε οικονομικό επίπεδο έχουμε παλιδρόμηση και υποθηκεύουμε το μέλλον τη χώρα μα δυστυχώ στο βάθρο τη εμπιστοσύνη των αγορών. Εξαιτία τη εμπιστοσύνη που θέλουμε να κερδίσουμε από τι αγορέ, υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μα. Και στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, δυστυχώς η Ευρώπη είναι μια τραγική απόδειξη παταγώδους αποτυχίας. Δυστυχώ δεν ε, καθοδηγούμε εμεί την παγκοσμιοποίηση, καθοδηγούμαστε από τις αγορές και δεν έχουμε εθνικές ε, κυριαρχίες πια. Έχουμε μόνο την κυριαρχία των αγορών. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το θέαμα. Ολόκληρε χώρες να καθοδηγούνται από τις δυναμικές τη αγορές και να χάνουν τους δικούς τους στόχου. Έτσι δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής και των πολιτικών. Και δυστυχώς δημιουργείται ένα δηλητηριώδες ε, κλίμα που ευνοούν τις εξτρεμιστικές δυνάμεις την άκρα δεξιά. Και δυστυχώς η δική μας απάντηση που χάθηκε μέχρι στιγμής είναι σαφής και επαναφέρει πυγμή και ε, δύναμη σε άλλες δυνάμεις που είναι ανώτερες, που δεν ε, υπόκεινται ε, στη λογική μόνο της αγοράς. Και αυτή η πυγμή, αυτό το σθένος ε, δυστυχώς της ε, άκρης δεξιάς εκμεταλλεύτηκε αυτή την δυσμενή κατάσταση και δυστυχώς θα έχει μεγάλη επιτυχία στις επόμενες ευρωεκλογέ και θα υπονομεύσει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Οπότε έχουμε δύο ερωτήσεις εδώ. Γιατί έχουμε μια τέτοια έξαρση της ακροδεξιάς. Είναι η απόδειξη της παταγόδους αποτυχίας των ε, διακρατικών δομών. Έτσι υποθηκεύσαμε και την κυριαρχία μας και υποτάξαμε τις δημοκρατικές δυνάμεις στην δυναμική των αγορών και ιδιαίτερα των χρηματοπιστών αγορών. Και μάλιστα ένα τμήμα της ε, Υπήρου μας δυστυχώς ε, υπέκυψε στις δυνάμεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και δυστυχώς αυτή την εμπιστοσύνη μόνο προσπαθήσαμε να κτίσουμε και όχι την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ε, Επόμενος ε, ο μιλητής, η κυρία Κρατιού. Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κάρας, ε, θα ήθελα να ευχαριστώ εσάς, ε, τον Μιχελάνχελ, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση της σημερινή συνάντησης. Χαίρομαι που ε, βρίσκομαι και πάλι εδώ, αυτή τη στιγμή εκπροσωπώντας τη γερουσία της Ρουμανίας. Θα ήθελα να πω κάτι που έχει σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Ρουμανία. Κοιτάξτε, ο απεσιόδοξος είναι απλά ένας ε, καλά ενημερωμένος ε, αισιόδοξο. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε σωστά ενημερωμένοι και αισιόδοξοι θα πρέπει να ομολογήσουμε παρόλα αυτά ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Πολλοί οργανισμοί ε, Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οργανισμοί, αλλά πολύ λίγες πολιτικές καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για να επιληθούν ε, τα ε, δημόσια, τα κοινά θέματα. Πράγματι υπάρχουν ε, δίκτυα, αλλά οι παγκόσμιοι θεσμοί αποδυναμώνονται όλο και περισσότερο τα Ηνωμένα Έθνη, η κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αντιμετωπίζεται πλέον, τουλάχιστον στο Βορρά, ως ένας τέτοιος θεσμός. Το θέμα που επιλέξαμε για σήμερα δείχνει ότι δεν αισθανόμαστε καλά με τη μη νομιμοποίηση αυτής της παγκόσμιας δράσης ή την αδύναμη νομοποίηση αν θέλετε. Νομίζω λοιπόν ότι τα κοινοβουλία έχουν εμπλακεί ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Αφενός έχουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς, τους οικονομικούς παίκτες ε, που εμπλέκονται σε διάφορες διαδικασίες για να επιλύσουν παγκόσμια οικονομικά προβλήματα και επιθυμούν να μην έχουν κανένα έλεγχο ή τουλάχιστον να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα κοινοβούλια. Και εν πάση περιπτώσει όταν πρόκειται για άτυπα δίκτυα ε, Πράγματι αυτό μοιάζει να είναι μία κοινή ιδέα. Από την άλλη βλέπουμε να αναδύονται νέα κινήματα της ε, συμμετοχικής ε, δημοκρατίας. Δυστυχώς λοιπόν αυτά τα κινήματα δεν μας ε, θεωρούν ικανούς τους εκπροσώπους για να περαπινθούμε των δημόσιων αγαθών μοιάζει να μην υπάρχει πλέον καθόλου χώρος για τα παλιά κοινοβούλια, αλλά πρέπει να υπάρχει τέτοιος χώρος. Η καλή διακυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν είναι δημοκρατική. Η οικονομική δύναμη μπορεί να ε, υπονομεύσει την δημοκρατία. Οι πολίτες αισθάνονται αντί ότι να ζουν σε κοινωνία, ότι ζουν σε μία αγορά. Νομίζω ότι ο Στίγκλιτς έχει δίκαιο που ισχυρίζεται ότι οι λειτουργίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικές όσο σήμερα. Όμως και ποτέ δεν υπήρχε τόσο περιορισμένη εμπιστοσύνη. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα που θέλω να θέσω. Θα μπορούσαμε άραγε να ιδρύσουμε μια παγκόσμια δημοκρατική διακυβέρνηση χωρίς να έχουμε ορίσει τι είναι τα παγκόσμια κοινά αγαθά και να έχουμε συντάξει τουλάχιστον κάτι γραπτό για να μπορέσουμε να υπεραμεινθούμε αυτών των αγαθών. Γνωρίζουμε ότι οι οικολόγοι κατόρθωσαν να προάγουν, να προστατεύσουν τη φύση και το περιβάλλον ως ένα δημόσιο αγαθό. Αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσει μας καθοδόν έχασαν την ειρήνη ως ένα δημόσιο αγαθό. Έχω και άλλες ερωτήσεις, τις φιλάω για αργότερα για το επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάινεν έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητέ Ότμα Κάρας και κύριε Μαρτίνες, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πραγματικά σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Τζόνσον και εγώ πριν από 40 χρόνια σπουδάσαμε στις Μπρουζ, στο Κολέγιο Ευρώπης, σπουδάσαμε και οι δυο μας διεθνή πολιτική και έκτοτε προφανώς και ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πολύ φίλε μου για τη δουλειά σου που ήταν πολύ σημαντική. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία ε, σε διεθνές επίπεδο, αυτό είναι το θέμα σου και πώς θα προαχθεί αυτή η δημοκρατία. Περνάμε λοιπόν στη συνεργασία ε, Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό σε μια εποχή της δυναμικής παγκοσμιοποίησης. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ καλούμεθα να υπεραμεινθούμε κοινών αξιών ε, σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Τα επόμενα χρόνια και τις ε, δεκαετίες ε, θα δούμε ότι θα ξετυλιχθεί μια συζήτηση για τις αξίες παράλληλα με πολλά άλλα θέματα. Εμείς η Ευρώπη ανάγουμε τον πολιτισμό μας από τις αξίες αυτές και ως πολίτες μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κοινά αγαθά ο 21ος αιώνας θα είναι τελείως διαφορετικός από το 19ο όταν ιδρύθηκε η IPU και ο προηγούμενος αιώνας επίσης. Με το διαδίκτυο πλέον έχουμε εντυπωσιακέ δυνατότητες αλλά έχουν προκληθεί και εντυπωσιακά προβλήματα. Αυτή η ιστορία με, τις, με την NSA της, των ΗΠΑ δείχνει ότι οι πληροφορίες μας και τα δεδομένα μας δεν ανήκουν πλέον σε εμάς αλλά σε κάποιες εταιρείες ή αν θέλετε σε κάποια κράτη. Αυτό λοιπόν είναι επίθεση κατά ε, θεμελιώδους δικαιώματος, ε, το οποίο είναι κατοχυρωμένο στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προφανώς και αναφέρομαι στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Το διαδίκτυο βέβαια έχει και την εκπληκτική δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα 7 δισεκατομμύρια πολίτες του κόσμου. Έτσι λοιπόν η διεθνής πολιτική δεν είναι ε, αποκλειστικό προνόμιο των κυβερνήσεων. Δεν ανήκει πια στις κυβερνήσεις αλλά στους ανθρώπους και υπάρχουν πολλές ε, παγκόσμιες κινήσεις ε, πολιτών με καλές προθέσεις και με πολύ καλή εξέλιξη. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας γνωρίζουμε ότι κυρίαρχος είναι ο πολίτης. Κατόπιν τούτου με ε, την κυριαρχία θα διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό κόσμο. Αυτό το στοιχείο της ε, κυριαρχίας είναι καθοριστικό στα κοινοβούλια. Όμως γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αυτοί που κινούν τα ενία της πολιτικής και δημιουργούν τα προβλήματα, κατ' ουσίαν είναι η τεχνολογία, το χρήμα που ρέει άφθονο στον κόσμο. Είδαμε τι συνέβη με την ε, οικονομική κρίση. Βλέπουμε ότι οι τράπεζες, τα hedge funds, αυτοί κατ' ουσίαν κινούν τον κόσμο και την οικονομία. Άλλος καθοριστικός παράγων είναι το διαδίκτυο, η φτώχεια και δυστυχώς σε κάποια μέρη του κόσμου η θρησκεία. Η θρησκεία η οποία καθορίζει και την πολιτική. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε την πρώτο καθεδρία της ε, πολιτικής ε, στην Ήπειρό μας, ε, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Και νομίζω ότι δεν τίθεται αμφιβολία από αυτού. Χρειαζόμαστε πιο έντονες προσπάθειες εκ μέρους των κοινοβουλίων για να μπορούν τα κοινοβούλια να διαδραματίσουν ρόλο. Από τη σημερινή μας συνάντηση ε, πρέπει να προκύψει το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό ε, η κάθε χώρα που έχει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίζεται με εμά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια για προτεραιότητες που έχουν πάρα πολλά ε, διεθνή φόρουμ. Μπορούμε από κοινού αν θέλετε να προγραμματίσουμε θεματολόγια, χρονοδιαγράμματα, θέματα. Ο κ. Τζόνσον ε, έδειξε ότι τελικά έχουμε πιάσει σχέσεις και με τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι εντυπωσιακό. Σε τελική ανάλυση τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός και ελπίζω να εξελιχθεί περαιτέρω. Ε, αυτά λοιπόν τα παγκόσμια αγαθά ε, μπορούν να τύχουν σωστή μεταχείριση σε τελική ανάλυση μόνο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι λιγάκι πιο φιλόδοξο. Θαυμάσιο το ότι έχουμε επιτύχει τόσα πολλά, αλλά σκεπτόμενοι το μέλλον πιστεύω δεν αρκούν αυτά. Εμείς έχουμε καθεστώς παρατηρητή. Και ισχύει και για άλλους αυτό. Και ο κύριος Τζόνσον είπε ότι ε, τα κοινοβούλια ε, εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα Έθνη, εμείς όμως δυστυχώς είμαστε παραπέδι των Ηνωμένων Εθνών. Ναι, μεν παριστάμεθα, αλλά δεν έχουμε άποψη και θεωρώ ότι η δημοκρατία θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να σκέφτεται και πιο πέρα και να μην ικανοποιείται με το ότι υπάρχει η Γενική Συνέλευση της Εκτελεστικής Εξουσίας, να διεκδικήσουμε Γενική Συνέλευση των Κοινοβουλίων. Στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχουν ε, εθνικά κοινοβούλια, αλλά ε, ευτυχώς ε, το 49 στο Συμβούλιο της Ευρώπης αποκτήσαμε κοινοβουλευτική συνέλευση. Άρα δηλαδή αν θέλει κανείς κάτι μπορεί να το επιτύχει. Και νομίζω ότι τα προβλήματα του κόσμου μας ε, οθούν στο να διεκδικήσουμε αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση και σε επίπεδο ΗΕ. Και θα επανέλθω στο θέμα αυτό το απόγευμα. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν πολλά και διαφορετικά θέματα και προβλήματα και νομίζω ότι καλό είναι όχι μόνο να θίγονται προβλήματα αλλά να κατατίθενται και προτάσεις. Δηλαδή τελικά τον καλύτερο συντονισμό πώς μπορούμε να τον επιτύχουμε. Ο κύριος Καϊνίντς από τη Λετωνία είναι ο επόμενος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω στα σχόλια που ακούσαμε στην αρχή για χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Νομίζω ότι πολύ σωστά αναφερθήκατε στην απογοήτευση και για την προσπάθεια και τις δραστηριότητες της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά το θέμα είναι και έλλειψη κατανόησης για το τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι κάνει και τι δεν κάνει σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. Ο εκλογέας δεν καταλαβαίνει πώς επηρεάζει τη ζωή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι κάνει διαφορετικά από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα μέσα ενημέρωσης συγκεντρώνουν την προσοχή τους στα αρνητικά της προσπάθειας αυτής και για πάρα πολλούς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μόνο στις Βρυξέλλες, είναι αποκομμένο από τον πραγματικό κόσμο. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Λετωνίας και με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης τέθηκαν πολλές ερωτήσεις για το πώς αυτή η νέα υπηρεσία θα συμπληρώσει και θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Τον τελευταίο χρόνο η Λέβη Άστον απέδειξε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει έναν ρόλο να παίξει. Επιτυχία στο Κωσίφο-Πέδιο, θετικότατος ρόλος στο Ιράν δείχνουν ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μπορεί να προσθέσει αξία στις εθνικές εξωτερικές πολιτικές. Εμείς μόλις μπήκαμε στην Ευρωζώνη σαν χώρα και η διαδικασία προς το ευρώ ήταν ομαλή, τίθενται θέματα βέβαια τώρα εκχώρησης αρμοδιοτήτων, τίθενται το θέμα της σχέσης της Ευρωζώνης με τη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Η αντιπαράθεση λοιπόν του εθνικού στοιχείου με, την ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό στοιχείο είναι κάτι που επανέρχεται συνεχώς. Τώρα για τον τίτλο αυτής της συνάντησης ε, «Παγκόσμια διακυβέρνηση και ε, κοινοβούλια». Η φράση «παγκόσμια διακυβέρνηση» «σφαιρική διακυβέρνηση» είναι κάτι που φοβίζει γιατί είναι κάτι που λειτουργεί απειλητικά για τα κράτη-μέλη, για τις χώρες γενικότερα. Πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια όπως λέγεται αλλά να δρούμε τοπικά και νομίζω ότι αυτό που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να βοηθήσει τη ζωή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια πρόκληση μπροστά μας και για τα Εθνικά Κοινοβούλια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπαιδεύσουμε σωστά τους συμπολίτε μας για το τι συμβαίνει εδώ στις Βρυξέλλες και πώς επηρεάζει τη ζωή μας. και πώς ταυτόχρονα δημιουργεί και κάποια θέματα περιορίζοντας λίγο αυτά που θέλουν να κάνουν. Αν θέλουμε λοιπόν να αυξήσουμε τη συμμετοχή των εκλογέων προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αποδεύσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στα μέλη του Προεδρείου, στους συναδέλφους ευρωβουλευτές και στους ε, ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η εισαγωγή της συνθήκης Λισαβόνας και η θέσπιση της τροποποίησε απότομα την ισορροπία δυνάμεων στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και ενώ οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξισορροπήθηκαν, διαπιστώθηκε μία διακρατικοποίηση, διακυβερνητικοποίηση και ενίσχυση, υπερβολική ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα διευθυντήριο στους κόλπους του Συμβουλίου. Κάτι που ήρθε σε αντίθεση ε, με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων που φαίνεται ότι έμειναν αγκιστρωμένα σε μια πολύ σημαντική μεν λειτουργία, αλλά ανεπαρκή, που είναι απλώς ε, ο έλεγχος ε, των εθνικών κυβερνήσεων. Και αυτή η ενίσχυση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου έδειξε κατάφορα το πόσο διαφορετική είναι η δύναμη επιρροής των διαφόρων χωρών στις λήψεις των αποφάσεων. Δημιουργήθηκε, παραλαμβάνω, ένα διευθυντήριο στο Συμβούλιο που, ε, κατά τη γνώμη των Ευρωπαίων, είναι ουσιαστικά η... το μόνο όργανο που λαμβάνει τις αποφάσεις, κάτι που διαταράσει την διαφάνεια και την δημοκρατική διαδικασία της λήψης των αποφάσεων. Και μάλιστα μερικές φορές οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τον ρόλο των κοινοβουλίων ε, καθόλου σημαντικό και αποφασιστικό γιατί φαίνεται ότι δίνουμε την εντύπωση ότι μιλάμε πολύ όταν μιλάμε αλλά ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει έμπρακτες συνέπειες και από τη στιγμή που δεν έχει έμπρακτη εφαρμογή και συνέπειες ε, δεν προβάλλεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άρα δεν φτάνει στους πολίτες. Εμείς γνωρίζαμε ότι με 28 χώρες ε, θα ήταν απαραίτητη μια μεταβλητή γεωμετρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι και διαφορετικές ταχύτητες, γιατί επιτράπηκαν κάποιες στρατηγικές ε, ε, κατασταλτικές που μερικές χώρες δεν αντιληφθήκαν ότι ήταν στρατηγικές αυτομαστίγωσης. Ήταν στρατηγικές κύρωσης ουσιαστικά σε επίπεδα ένωσης που μετατρέπονται σε στρατηγικές αυτομαστίγωσης της ίδιας της ένωσης. Η ερώτηση όμως που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι πώς θα εγκύψουμε στο θέμα αυτό. Φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, πρέπει να καταφέρουμε αυτά τα Εθνικά Κοινοβούλια να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά να δίνουν και ισχύ και δύναμη στις εθνικές κυβερνήσεις για να έχουν επιρροή στη διαμόρφωση των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και να ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω πάντως, όπως είπε και ο Σέρζιο Σόουζα Πίντο, ο πρώτος ομιλητής, είναι κάτι που δεν θα πρέπει, είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Το πώς ε, αξιολογούν οι Ευρωπαίοι πολίτε, και εξού και η μεγάλη αποχή, το, την πραγματική εξουσία των ε, θεσμικών οργάνων. Όλο και περισσότερο οι Πορτογάλοι αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα είναι εχμάλωτα, είναι όμοιροι και μάλιστα θεωρούν ότι είναι εχμάλωτα αυτά τα όργανα στην σε μια πρακτική που δεν είναι πάντα δημοκρατική παρόλο που είναι δημοκρατικές εκλογέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρισκόμαστε κατά τη γνώμη σε, μια, σε ένα σημείο καμπή. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την πολιτική και αλληλέγγυα διάσταση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών και την πίστη του στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Ευχαριστώ. Äh, ο επόμενο ομιλητή είναι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κύριο Μουσουρούλη, παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι η κρίση έχει αλλάξει τον τρόπο που οι λαοί μας αντιλαμβάνονται τα πράγματα, σκέφτονται, δρούν και αντιδρούν. Και ασφαλώς αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαση την πολιτική τάξη, η οποία πολλές φορές έδειξε ότι καθοδηγείται από την οικονομία, από την αγορά, ε, καλώντας και τα εθνικά κοινοβούλια στην ουσία να περάσουν σε μια προσαρμογή ε, οικονομικών αποφάσεων σε μια πολιτικοποίηση αν θέλουμε ε, ε, οικονομικών αποφάσεων. Είναι επίσης αλήθεια ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το βάρος της κρίσης το σήκωσαν τα εθνικά κοινοβούλια και των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα αλλά βεβαίως και των χωρών που στήριξαν αυτό το πρόγραμμα. Αυτό, ξέρετε, αναβίωσε τις παραδοσιακές διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ πληρωτών καθαρών πληρωτών και λιπτών, οι οποίες υποκαταστάθηκαν από τις νέες σχέσεις μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών. Ε, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε σε πολιτικό επίπεδο, οριακές πλειοψηφίες, ε, τριγμή στη συνοχή των κοινοβουλευτικών ομάδων και βέβαια αρνητική φόρτιση και στις δύο περιπτώσεις της κοινή γνώμης. Ε, αυτό είναι το τοπίο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, ως αιρετή στις επόμενες εκλογές. Διέγνωσα ότι μία, μία και μόνο κίνηση, δηλαδή η συγκρότηση της Επιτροπής Κάρας για το θέμα της, του τρόπου λειτουργίας της ε, Τρόικα, αντιστάθμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αρνητική προδιάθεση της κοινή νόμης απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με μία μόνο κίνηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την, ε, την χώρα μου, την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, σημείωσα μάλιστα, νομίζω εσείς το είπατε, ότι όσα περισσότερα γνωρίζει ο πολίτης για την Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η προσέλευση στις εκλογές. Ε, επιτρέψτε μου να βάλω ένα ερωτηματικό. Μπορεί να έρθει στι ευρωεκλογέ, αλλά για να καταψηφίσει την Ευρώπη, όχι για την υπερψηφίσει. Άρα λοιπόν πρέπει, ε, ε, να βρούμε και άλλου τρόπου να περάσουμε θετικά μηνύματα. Τώρα, ε, είναι αλήθεια ότι έχουμε μία καταγεγραμμένη επιστροφή στον εθνοκεντρισμό. Και το παράδοξο εδώ, το είπα και χθε στο δίκτυο που έχουμε το Ευρωπαϊκό Λογικό Κόμμα, το παράδοξο εδώ είναι ότι αυτή την επιστροφή τη βλέπουμε και σε χώρες που δεν έχουν ε, προβλήματα από τις επιπτώσεις κρίσης. Παράδειγμα, Ελβετία με ανεργία 3,2%, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κλπ. Αυτή λοιπόν ε, η, η μεταστροφή των, λαών ε, στις, στα εθνικά κράτη αλλά και στις, στα κράτη όπου υφίσταται έντονα τις επιπτώσεις κρίσης η αποστροφή των πολιτών λόγω της απόγνωσης που δημιουργεί η κρίση από τη δημοκρατία, εξού και η άνοδος της ε, άκρας δεξιάς, επιβαρύνουν πολύ το πολιτικό τοπίο. Συνεπώς, για να, για να ε, κλείσω αυτή την, ε, την παρέμβαση, δεν υπάρχει ερώτημα. Αν θα μπορούσε να δημορφωθεί και ένα ερώτημα, δηλαδή τι είναι αυτές οι, οι θετικές πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει το Ευρωκοινοβούλιο, όπως η Επιτροπή Κάρας, που θα έχουν θετική απήχηση στους ευρωπαϊκούς λαούς και πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς ελέγχου ad hoc, ad hoc ε, δομών, όπως για παράδειγμα η Τρόικα, θνησιγενών αν μου επιτρέπετε, διότι ε, δεν, ε, ο ρόλος τους έχει ήδη υποκατασταθεί από θεσμικό πλαίσιο, από κανονιστικό πλαίσιο, συγκεκριμένα τον κανονισμό 472, ο οποίος οργανώνει την εποπτεία των χωρών ε, που έχουν πρόβλημα χρέους. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα τελειώσει και βεβαίως μηχανισμοί ελέγχου άτυπων συνελεύσεων ε, και άλλων ε, διεθνών φόρουμ όπου λαμβάνονται πολύ ισχυρές αποφάσεις που καλούμαστε εμείς να ενσωματώσουμε στη συνέχεια μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία χωρίς όμως να υπάρχει πραγματικά ουσιαστικός έλεγχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά να προβληματιστούμε ε, στο θέμα αυτών των, των, πρωτοβουλειών. Ε, και το λέω αυτό και το τονίζω ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τι, τι απήχηση είχε στην Πορτογαλία ή στην Ιρλανδία ή σε άλλες χώρες κρίσης, αλλά με μία μόνο κίνηση άλλαξε η εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you uh, από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, ο κ. Μέρφυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα. Συνεχίζοντας αυτά που έλεγε ο Έλληνας φίλος και συνάδελφος Συζητάμε για τη δημοκρατία, για τη συμμετοχή και ο κύριος Μαρτίνες αναφέρθηκα στα προβλήματα που νιώθει ο κόσμος και αυτό μετατρέπεται σε χαμηλή συμμετοχή. Το βασικό κίνητρο για τον κόσμο να πάει να ψηφίσει είναι αν θεωρεί ότι έχει σημασία αυτό το οποίο θα κάνει. Σαν παράδειγμα, η υψηλότερη συμμετοχή που είχαμε σε γενικές εκλογές ε, εδώ και τρία χρόνια έγινε μόλις είχαμε μπει στη δική μας διαδικασία bailout. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το δημοψήφισμα που είχαμε κάνει για το Σύμφωνο Σταθερότητας Δημοσιονομικής. Τα πράγματα μπορεί στην Ιρλανδία να τα βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα ή κάποιες άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, ο λαός σε σχέση με την Τρόικα δεν είχε να πει τίποτα, αλλά μερικούς μήνες μετά του τέθηκε το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας. Γνωρίζω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δική μου χώρα είχε υπάρξει μια ελπίδα για να μην υπάρξει δημοψήφισμα, αλλά στο δημοψήφισμα το 60% στήριξε το σύμφωνο και υποστήριξε ουσιαστικά τους όρους της Τρόικα και του Bailout. Έτσι λοιπόν οι πολίτες θεώρησαν ότι ελέγχουν οι ίδιοι ότι συμμετέχουν στη διαδικασία του Bailout. Υπήρξε φυσικά ιδιαίτερη εμπλοκή και των κοινωνικών εταίρων και υπήρξαν πολλές ισχυρές αντιπαραθέσεις. Αλλά ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση την οποία έπρεπε να πάρουμε, η πιο δύσκολη ίσως από το 1920 που δημιουργηθήκαμε. Χαμηλή συμμετοχή για τις ευρωεκλογές όμως, αλλά ο λόγος είναι η σημασία που δίνει ε, ο πολίτης σε αυτό το οποίο κάνει το κοινοβούλιο. Ήμουνα εδώ και δύο εβδομάδες στην διακοινοβουλευτική συνάντηση σε αυτήν εδώ την αίθουσα και πάρα πολλοί πήραν το λόγο από διάφορες χώρες και από πολλά πολιτικά κόμματα. Στο τέλος της συζήτησης δεν υπήρξε κάποια απόφαση, δεν υπήρξε κάποια προσπάθεια να υπάρξει μια κοινή απόφαση. Αν εμείς αναπτύξουμε τη διακοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα να γίνει ένα φόρουμ το οποίο να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να παίρνει αποφάσεις, να κάνει συστάσεις, τότε <clears throat> ε, οι πολίτες ε, δεν θα πρέπει να τους υποτιμάμε γιατί ξέρουν τι έχει σημασία. Δεν θα τους πούμε εμείς τι έχει σημασία. Εμείς θα πρέπει να καταστήσουμε τα θεσμικά όργανα σημαντικά. Για να το πετύχουμε αυτό ε, ξέρετε ότι εμείς στην Ιρλανδία θα έχουμε την ίδια μέρα τοπικές, δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Όταν ψηφίζουν λοιπόν για ευρωεκλογές, ε, οι πολίτες ουσιαστικά ψηφίζουν τις επιδόσεις ε, της κυβέρνησής τους. Επίσης ψηφίζουν σε πολιτικό επίπεδο, αν είναι σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες ή κάτι άλλο. Και ένα μικρό τμήμα μόνο του κινήτρου ψηφοφορίας είναι τα όργανα της Ένωσης. γιατί πράγματι ο κόσμος ε, όταν ψηφίζει στις ευρωεκλογέ ναι μεν δεν φοράει την φανέλα της εθνικής του ομάδας αποκλειστικά αλλά σκέφτεται για τη ζωή του ο καθένας, πώς θα βελτιώσει τη ζωή του από την ψήφο του. Και αν είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες όλοι και περισσότερο θα ψηφίσουν. Πρέπει με απλό τρόπο να δείξουμε στον κόσμο γιατί πρέπει να ψηφίσει. Εμεί στην Ιρλανδία συζητάμε σαν παράδειγμα την πολιτική αγωγή στα σχολεία, να χαμηλώσουμε επίσης ε, το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στις εκλογές, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει ούτε πώς ψηφίζει, ούτε πού να ψηφίσει. Τέλος, αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω γιατί είμαι εδώ στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα είναι στην ίδια φάση με μένα. Αυτά σε ένα παγκοσμιημένο κόσμο πρέπει να διορθωθούν. Πολλοί από εμά ταξιδεύουν ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν σε άλλη χώρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σα ευχαριστώ. Τι εννοείτε, ένα παγκόσμιο σύστημα ψήφου ή εκλογικό. Ο κύριος Γκρέχ. Από τη Μάλτα. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Κάρα. Σας ευχαριστούμε και τη διοργάνωση αυτή τη συνάντησης. Θα ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Τζόνσον για την ε, παρουσίασή του και για τις ε, σκέψεις του για το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι τα σχόλιά του υποβάλλονται την ε, κατάλληλη χρονική στιγμή. Βέβαια, όπως ε, διαπιστώσαμε στις συζητήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί, ε, βλέπουμε πως η πολυμέρεια μπορεί να ενισχύσει το στόχο και το ρόλο των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό βέβαια μπορεί να καταστεί πρακτική εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία ξεκινάει από τη δημιουργία οικονομικής δύναμης αλλά και κοινωνικών εξελίξεων που εντάσσονται στο πλαίσιο των αξιών μας. Επίσης ε, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στο ότι υπάρχει το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης πλέον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι που το βιώνουμε στην ε, καθημερινή μας ε, ζωή. Κυρίως αυτό τον κόσμο που ε, υπάρχει ένα θεσμικό, μάλλον ψηφιακό πλαίσιο και όλες οι χώρες είναι συνεδεμένες μεταξύ τους. Για μένα, για τη Μάλτα, η παγκοσμιοποίηση ε, έχει πολύ σημαντικότερες επιπτώσεις ε, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα. Οι επιπτώσεις λοιπόν της πολυμέρειας σε αυτόν τον κόσμο της παγκοσμιοποίησης μας επηρεάζουν άμεσα ε, και αν θέλετε αναλογικά ε, επηρεαζόμαστε πολύ περισσότερο από άλλες χώρες και αυτό πάλι οφείλεται στο μέγεθος της χώρας μας όπως σας είπα. Κάτι άλλο ο τρόπος ε, με τον οποίο οι εθνικές συνελεύσεις μπορούν ε, να επηρεάσουν περισσότερο τη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να προβάλλω αυτό το στοιχείο της ε, σημασίας γιατί αν δεν υπάρχει ε, σημασία και ενδιαφέρον τότε δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη και αυτό σε τελική ανάλυση τελικά δηλαδή θα αφαιρέσει και από το λόγο ύπαρξης των κοινοβουλίων και των πολυεθνικών θεσμών. Πιστεύω λοιπόν ότι τελικά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αδιαφορία απέναντι στην πολιτική και θα οδηγήσουν και σε μικρότερη ε, συμμετοχή ε, στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε το, την κοινοβουλευτική διάσταση των πολυμερών αυτών ε, συνελέψεων χωρίς να αφαιρέσουμε από την ε, επικουρικότητα, χωρίς ε, να μειώσουμε τις νομοθετικές και διοικητικές αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Με πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αυτή η έννοια πάνω απ' όλα μπορεί να γεφυρώσει και να συγχωνέψει ε, τα πολιτικά θεματολόγια σε τρία διαφορετικά επίπεδα. το επίπεδο το πολυμερές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι αυτή η σύγκληση, αυτή η ευθυγράμμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει πλέον διαχωρισμός ανάμεσα σε προτεραιότητες που είναι σημαντικές για τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι ορισμένα θέματα που συζητούνται σε πολυμερείς συνδιασκέψεις δεν είναι απαραίτητα η προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα των πολιτών. Πάντως αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι ε, να επιδιώξουμε την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Και αυτή η σύγκληση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από, μια, από ένα πραγματικό θεματολόγιο. Τα θεματολόγια να είναι πραγματικά, ρεαλιστικά από οικονομική σκοπιά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή να είναι μια νέα πλατφόρμα όπου θα δώσουμε ε, πραγματικές απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, άλλους πέντε ομιλητές έχουμε αλλά νομίζω ότι παρόλα αυτά καλύτερα να δοθούν οι πρώτες απαντήσεις. Κύριε Τζόνσον, έχετε το λόγο. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να δώσω απαντήσεις, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση. Δια... Διαπίστωσα ότι πολλοί αναφερθήκατε στις προβλέψεις για πολύ χαμηλή προσέλευση στις κάλπες ε, και ε, όχι, ιδιαίτερη όχι ιδιαίτερα καλή γνώμη που έχουν οι πολίτες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε βουλευτής ε, στον κόσμο παρακολουθεί δημοσκοπήσεις, ε, συμμετρήσεις που γίνονται παντού και παντού τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Οι ε, κοινοβουλευτικοί θεσμοί, και τα μέλη αυτών των κοινοβουλευτικών θεσμών βρίσκονται, αν όχι στην τελευταία σειρά, στην τελευταία θέση, σίγουρα στις, στις τελευταίες θέσεις ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έγινε μία μελέτη γιατί ισχύει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι υπάρχει μία οικουμενική απάντηση. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί αυτή η εικόνα των πολιτών για τους πολιτικούς, αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι μοιραία και έχουν σχέση με την ίδια τη φύση της πολιτικής. Όταν κανείς κατεβαίνει σε εκλογική εκστρατεία, το κάνει για να κερδίσει ψήφους. Έχει ένα πρόγραμμα, ένα εκλογικό πρόγραμμα και δίνει υποσχέσεις ε, ότι θα υλοποιήσει συγκεκριμένους στόχους. Και είναι στη φύση των πραγμάτων ότι δεν θα καταφέρετε να τους υλοποιήσετε αυτούς τους στόχους. Οπότε, αν χρόνο με το χρόνο υποσχόμαστε στους πολίτες ότι θα επιφέρουμε κάποιες αλλαγές και διαπιστώνει οι πολίτες ότι δεν είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να κρίνουν οι πολίτες ότι δεν είμαστε και πολύ σοβαροί, μια και δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να σκεφτούμε είναι ποιο είναι το μήνυμα που δίνουμε στους πολίτες. Και γι' αυτό θα αναφερθώ στο θέμα της σημασίας ε, και του βάρους. Τι βάρος και πόσο σημαντική, τι έχουμε και πόσο σημαντικοί είμαστε για τους πολίτες. Πριν από κάνα δύο χρόνια ολοκληρώσαμε ένα διετές πρόγραμμα στο οποίο κάναμε ε, δημοσκοπήσεις ε, για τη γνώμη των πολιτών και τη γνώμη των βουλευτών για τη σχέση μεταξύ τους. Και διαπιστώσαμε ότι ισχύει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι πολίτες ρωτούσαν τους βουλευτές τι κάνετε για μας, δεν ενδιαφέρει τους πολίτες τι κάνουν οι βουλευτές για την γενική κατεύθυνση, την πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι τι κάνει ο ΑΒ βουλευτής για τον πολίτη. Γιατί ο πολίτης ε, θέλει δουλειά, θέλει ε, παιδεία για τα παιδιά του. Τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Και αυτό θέλει ο πολίτης, αυτό περιμένει από τον ε, πολιτικό που εξέλεξε από το βουλευτή. Ενώ οι βουλευτές θεωρούν ότι όλο και περισσότερο χρόνο του κοινοβουλευτικού του έργου το αφιερώνουν στην προσπάθεια της ε, να ικανοποιήσουν τις ανησυχίες των ε, εκλογέων τους. Αυτό πιστεύουν οι πολιτικοί και οι βουλευτές ότι κάνουν ό,τι μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ε, συμπολίτες τους, αλλά φυσικά υπάρχουν όρια σε αυτό, στο τι μπορεί να κάνει κάθε βουλευτής. Πάντως, ε, πολλά κοινοβουλία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την ιδέα ότι είναι απόντες από τη ζωή των πολιτών είναι να κάνουν τα κοινοβουλευτικά τους όργανα πιο διαφανή, ώστε να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν με εύκολο και προσιτό τρόπο τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι τρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι τρέχει στην ε, Εθνική Βουλή και επίσης ε, να μπορεί ο πολίτης να δίνει κάποιο input σε αυτό που συμβαίνει στο κοινοβουλευτικό έργο. Βέβαια, μερικέ χώρες έφτασαν στα άκρα. Μπορεί κανεί ε, μέσω του διαδικτύου ή με άλλα μέσα ένας πολίτης να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση συγκεκριμένων ε, νομοθετικών διατάξεων. Και έχουμε πολυμελή προσωπικό που επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία, τις συνεισφορές ουσιαστικά των πολιτών και το τι περιμένουν από την νομοθεσία. Το διαδίκτυο και οι τεχνολογίες της ε, πληροφορίας μας δίνουν τεράστιες ευκαιρίες ε, ώστε να συμπεριλάβουμε και τις απόψεις των συμπολιτών μας στο νομοθετικό έργο. Πάντως ε, έτσι πιστεύω ότι θα αποκτήσει και το κοινοβουλευτικό έργο μεγαλύτερη σημασία και θα έχει και μεγαλύτερο βάρος στα μάτια του πολίτη. Τώρα, είδαμε και την αντιπαράθεση της παγκόσμιας διάστασης με την εθνική διάσταση. Και είπαμε ότι θα πρέπει να αποκαταστήσουμε περισσότερη δημοκρατία στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι αναφυσβήτητο, ότι όλοι μιλούμε για το ίδιο πράγμα και επιδιώκουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχει, υπάρχει μια τεράστια αντίσταση και δεν μας άρεσε το λόγο, τεράστια αντίσταση σε αυτό. Γιατί για αιώνες ολόκληρους ε, ε, αυτή ήταν η μορφή συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Και θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Το 2005 πήγα με μια ομάδα Προέδρων Βουλών στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη και είχαμε μια ενημερωτική συνάντηση με τους πρέσβεις για αυτή τη διάσκεψη των Προέδρων Βουλών που θα γινόταν αργότερα με συνόδευε ένα πρόεδρο Βουλή που μάλιστα αυτή τη στιγμή είναι και πρόεδρο στη χώρα του, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καθόταν δίπλα μου λοιπόν και κάνω αυτή την ενημέρωση στου πρέσβει για το τι θα συζητούσαμε, για τη σημασία που έχει μια τέτοια συνδιάσκεψη και τον απότερο στόχο να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη δημοκρατία στα Ηνωμένα Έθνη. Κατά το τέλος της συζήτησης, ένας πρέσβης ε, συμπατριώτης μάλιστα του Προέδρου που ήταν παρακαθημένος μου, είπε «Φυσικά είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, σας υποδεχόμαστε με ανοιχτέ αγκάλες, στο μέτρο όμως που λέτε τα ίδια με αυτά που λέμε κι εμείς». Και νομίζω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης, ότι υπάρχει διακρατικός θεσμός, διακρατική συνεργασία και οι χώρες δεν θέλουν τέτοια αλλαγή προς περισσότερη δημοκρατία δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο σύντομα τουλάχιστον. Γι' αυτό θα το πρέπει να το κάνουμε σταδιακά, βαθμιδών. Δηλαδή να φέρουμε τα κοινοβούλια πιο κοντά στα Ηνωμένα Έθνη. Να συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότερο στι διαδικασίε. Και αν θέλετε να συμμετέχετε στι συζητήσει για τη δημιουργία τη ειρήνη, υπάρχει ειδική επιτροπή στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορείτε να πάτε εκεί. Το ίδιο γίνεται και στο Συμβούλιο για τα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πήγα προχθέ στην Ρουμανία και είχαμε συνάντηση με 12 βουλές και συζητήσαμε το πώς μπορούν αυτές οι βουλές να λαμβάνουν μέρος στην ε, ετήσια ε, παγκόσμια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν συμμετοχής. Υπάρχουν ήδη πολλοί άριθμοι τρόποι συμμετοχής. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους τρόπους γιατί σε πολλές διαδικασίες υπάρχουν δυνατότητες να επηρεάσετε τις διαπραγματεύσεις σε όλα αυτά τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Äh, Πολύ ωραία. Πριν λοιπόν ε, ε, περάσουμε και σε άλλες απαντήσεις, καλύτερα να κάνετε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Ρικάρντο Μπατίστα από την Πορτογαλία. Bon Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στις Βρυξέλλες και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεται να κάνουμε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Σημαντική και για τις χώρες μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Φυσικά δεν μπορούμε να αγνοούμε τις διαστάσεις της της πορτογαλικής αντιπροσωπείας σήμερα σε αυτή τη συζήτηση και ο πρόεδρος ε, της Πορτογαλικής Βουλής θέλησε με την πολυμελή αυτή αντιπροσωπεία να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα της Πορτογαλίας στην διάσκεψη αυτή. Και το πρώτο μήνυμα είναι ότι έγιναν λάθη που δεν θα πρέπει να επαναληφθούν σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Κάρας είπε ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματα της κρίσης. Η αξιολόγηση της Τρόικας και του έργου της Τρόικας είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει. Και έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα με άμεση ψηφοφορία, αλλά παρόλα αυτά δεν αποφεύθηκαν κολοσσία λάθη ε, στη διαμόρφωση του μνημονίου που οδήγησε σε μια πολύ κακή κατάσταση στην Πορτογαλία γιατί δυστυχώς ε, ε, είχαμε πολύ κακή εκτίμηση, ανακριβή εκτίμηση του ελλείμματος με ολέθρια αποτελέσματα. Στην υγεία επίσης επικεντρωθήκατε μόνο στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα και δυστυχώς ε, καταλήψατε όλα τα θέματα δημόσιας υγείας που είναι πολύ σημαντικά και επίσης ε, δεν ε, εγκρίθηκαν μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της χρηματοπιστωτικής παρέμβασης που έγινε στην Πορτογαλία και του προγράμματος διάσωσης. Και πολλές φορές ε, ακούσαμε ε, εκπροσώπους της Τρόικα να βρίσκονται στο πλευρό του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου και να λένε ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να είναι μια οικονομία με χαμηλό α, ε, κόστος εργασίας. Δεν είναι αυτός ο δρόμος της Πορτογαλίας, ούτε θα μπορούσε να είναι αυτός ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ταυτόχρονα λένε ότι δεν επηρεάζεται την κυριαρχία του κράτους μέλους. Οπότε, αν τα εθνικά κοινοβούλια είχαν αναμειχθεί σε αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων που έχουν σημαντική επιρροή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσω θα είχαμε αποφύγει κάποια τέτοια λάθη. Κύριε Τζόνσον, είστε Γενικό Γραμματέα τη ε, Διακοινοβουλευτική Ένωση και σα συγχαίρω για τα 125 χρόνια ζωή του θεσμικού σα Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα και η συμμετοχή τη ε, IPU. Γιατί θέλουμε ένα πιο ενεργό ρόλο των ε, κοινοβουλίων στου διεθνεί οργανισμού. Είναι αλήθεια ότι εμείς οι εθνικοί βουλευτές που εγκρίνουμε τους, εμείς εγκρίνουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς και εγκρίνουμε ουσιαστικά και τα κονδύλια που καταβάλουν οι χώρες μας στους διεθνείς οργανισμούς. Οπότε είναι απαραίτητο να συμμετέχουμε και εμείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει να ασκούμε έναν ουσιαστικό ρόλο. Επίσης, ε, ρόλος μας είναι να ελέγχουμε και τις επιλογές αυτών των ε, ε, διεθνών οργανισμών και των θεσμικών οργάνων, κάτι που δεν γίνεται πάντα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε το παρόν σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και οργανώσεις. Επίσης θα πρέπει και το πρόγραμμα αυτών των διεθνών οργανισμών να ευθυγραμμίζεται με το, τα ενδιαφέροντα των συμπολιτών μας. Να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα των πολιτών και να γίνονται σεβαστά τα παγκόσμια συμφέροντα, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Συμμετείχα πολλές φορές στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Και φαίνεται όλο και πιο καθαρά, όλο και περισσότερο, ότι οι επιλογές για τις επενδύσεις των οργανισμών αυτών εξαρτώνται περισσότερο από τους ε, βασικούς δωρητές, ε, από τους πραγματικούς συνεισφορείς και από τις δικές τους επιλογές και δεν ε, υπακούν οι επενδύσεις ε, στα πορίσματα των επιστημόνων ή στις ανάγκες που έχουμε για την υγεία ή για την ανάπτυξη. Μιλήσατε για τους στόχους μετά το 2015. Θα πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη των ασφαλμάτων του παρελθόντος και θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ε, εθνικούς βουλευτές που είναι οι άμεσα εκπρόσωποι των πολιτών και έχουν και την δημοκρατική νομιμοποίηση να τους επιτρέψουμε να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο του ρόλου και των δραστηριοτήτων των διεθνών οργανισμών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον πρώην Επίτροπο και νυν ε, βουλευτή από την Ουγγαρία, τον κύριο Κόβατς. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης και τον Μιγκουέλ Άγχελ και τον κύριο Κάρας για τις εισαγωγικές τους παρατηρήσεις και τέλος θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τζόνσον για την ιδιαίτερα ενημερωτική κεντρική του ομιλία. Το πιο έντονο χαρακτηριστικό της ε, καθημερινότητάς μας είναι η παγκοσμιοποίηση. Είναι μια αντικειμενική διαδικασία, είτε μας αρέσει ή όχι, η οποία δεν μπορεί να αναστραφεί ή να σταματήσει. Οι προκλήσεις όπως η αποκατάσταση της ειρήνης, η ασφάλεια, η σταθερότητα, η τρομοκρατία, η οικονομική κρίση, η έμβια, η λοιμή, οι επιδημίες είναι προβλήματα πλέον παγκόσμια. Οι παγκόσμιες προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθνικά μέτρα και σε ένα εθνικό πλαίσιο. Μπορούν να αντιμετωπιστούν όμως μέσω της διεθνούς διακυβέρνησης. Βασικός στόχος των κοινοβουλίων είναι ο νομοθετικός φυσικά, το να παράγουν νόμους. Ταυτόχρονα όμως τα κοινοβουλία ανήκουν στο σύστημα των ελέγχων, το checks and balances σύστημα. Είναι βασικό εργαλείο της δημοκρατίας. Εκπροσωπούν άμεσα τους εκλογίστους Εκπροσωπούν τις φιλοδοξίες, τις επιθυμίες, και τις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις στις χώρες τους. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών ανάμεσα στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις, οι σχέσεις του και η συνεργασία του σε εθνικό επίπεδο είναι πρότυπο, πρότυπο συγγνώμη, και για τις διακυβερνητικές και διακοινοβουλευτικές οργανώσεις. Τα εθνικά κοινοβούλια και οι διακοινοβουλευτικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση των διεθνών σχέσεων. Θεωρώ ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διακυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να ενθαρρύνουν τον κοινοβουλευτικό κλάδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ειδική κοινότητα που βασίζεται σε βασικές αρχές όπως το κράτος δικαίου, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δημοκρατία. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει η δυνατότητα να εκπληρώσει την αρμοδιότητά της η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Είναι μια περίπλοκη δομή αυτή που έχει, αλλά παρόλα αυτά οι αξίες της επιτρέπουν να παίξει σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Είναι ένα βασικό επιχείρημα για τη συμμετοχή σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις και ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Το θέμα ξέρω ότι εκρεμεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Σωστή διεθνής διακυβέρνηση πρέπει να εκπληρεί ορισμένα κριτήρια. Η διεθνής διακυβέρνηση πρέπει να είναι βασικά δημοκρατική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, μπορούν να δώσουν το παραδείγμα. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Πρώτον, η δραματική οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και 2009 που δεν έχει ακόμα τελειώσει. Είναι προϊόν της ε, έλλειψης δημοκρατικού ελέγχου στις διεθνείς αγορές. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερο θέμα, η Αραβική Άνοιξη. Τα αυταρχικά καθεστώτα που είχαν καλές σχετικά οικονομικές σχέσεις με κάποιες χώρες μέλη, κατέρευσαν με ξαφνικό τρόπο και μας έδωσαν ένα καλό παράδειγμα. Η πολιτική σταθερότητα στην επιφάνεια που βασίζεται σε αντιδημοκρατικές πολιτικές τελείωσε. Στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να δίδουν προτεραιότητα στις οικονομικές αξίες αλλά στις αξίες της δημοκρατίας. Και τρίτον, έχουμε ευρωεκλογές τον Μάιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών διαφορετικών πολιτικών οικογενειών θα πρέπει να διεξάγουν μια πολύ εντατική εκστρατεία για να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και να ελαχιστοποιήσουν τις επιρροές των ευρωσκεπτικιστών και των δυνάμεων εναντίον της Ευρώπης που είναι και εναντίον της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόβατς. Επόμενος είναι ο κύριος Πίμενοφς από τη Λετωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην ε, επιστολή που μας στείλατε πριν από τη συνάντηση, στην πρόσκλησή σας και εκεί επελαμβάνεται η ουσία του θέματος που συζητάμε. Η παγκόσμια διακυβέρνηση δεν πρέπει να παραμείνει μόνο στα χέρια των κυβερνήσεων και των ε, διπλωματών, αλλά πρέπει να αφαιθεί και στα κοινοβούλια, γιατί τα κοινοβούλια παίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτή η επιστολή υπογράφεται από τους κυρίους Κάρας και Μαρτίνες. Εγώ λοιπόν ισχυρίζομαι το εξής. Πριν ενισχύσουμε τα εθνικά κοινοβούλια, πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να αποκτήσουν περισσότερες αρμοδιότητες. Εάν το κοινοβούλιο είναι ο μικρός αδελφός μιας κυβέρνησης, τότε μπορεί να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο. Μπορούν τα κοινοβούλια να παρεμβαίνουν σε εθνικές υποθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των Εθνικών Κοινοβουλίων προσφέροντας ε, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται τα κοινοβούλια για να επηρεάζουν τις ε, αποφάσεις των κυβερνήσεων. Κυρίως σε θέματα που έχουν σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ε, σημαντικές αποφάσεις που είναι καθοριστικές ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορώ να σας ε, τεκμηριώσω αυτό μου το επιχείρημα. με την ένταξη της Λετωνίας στην Ευρωζώνη, κάτι που συνέβη πρόσφατα στις αρχές αυτού του έτους. Πέρυσι, την άνοιξη του 2013, Μόνο το 1 τρίτο των Λετωνών ήταν υπέρ της ε, υιοθέτηση του ευρώ στη Λετωνία. Το Δεκέμβρη ήταν 15% αλλά ή μάλλον 50% αλλά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Και έκτοτε στη δική μας ε, τη χώρα ε, δεν έχει κληθεί το Κοινοβούλιο να ελέγξει τελικά ποια είναι η βούληση του λαού. Είναι ο λαός υπέρ του ευρώ. Είναι υπέρ του, του να αφήσουμε το εθνικό μας νόμισμα για να υιοθετήσουμε το ευρώ. Και μόνο η κυβέρνηση ήταν αρμόδια για αυτή την απόφαση. Ξέρω, οι αντίπαλοι μου θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι κατά τα παλαιότερα έτη το Κοινοβούλιο μπορούσε να επηρεάσει αποφάσεις κυβέρνησης. Εδώ θέλω να υπογραμμίζω ότι αυτή η απόφαση ελήφθη μόνο από την κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, τι είδου ε, επιρροή μπορούμε να περιμένουμε από εθνικά κοινοβούλια, αν τα κοινοβούλια δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Οι βουλευτές μπορούν να λαμβάνουν σωστά τις αποφάσεις ε, αν δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και πιστεύω ότι αυτό που είναι απαραίτητο να υπάρχει είναι ένα σύστημα που να έχει άμεση σχέση με την παιδεία και την ενημέρωση των κοινοβουλίων πριν καλέσουμε τα κοινοβούλια να ε, συμμετάσχουν ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Νομίζω ότι Ίσως εδώ πολλοί στην αίθουσα πιστέψουν ότι το επιχείρημά μου είναι πολύ συντηρητικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι η ανάληψη ευθυνών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν και αυτά να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τζοζέ Μαγκάλες. From Portugal. Από την Πορτογαλία. Πολύ οι Πορτογάλοι σήμερα. Τι, τι αντιπροσωπεία είναι αυτή, πάρα πολύ ισχυρή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά που πολύ σωστά μας ε, παρουσίασε ο κ. Τζόνσον, δηλαδή τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί βελτιώνεται η συνεργασία και η ψηφιακή εποχή την ε, ευνοεί. Έχουμε δίκτυα κοινοβουλευτικά και όλο και περισσότερους βουλευτές που μπορούν να, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες Πραγματικά με εντυπωσιάζει πόσο εύκολη είναι πια η επαφή χάρη στην ε, πληροφορική. Για παράδειγμα στο Global Action όλη η ελογραφία γίνεται ηλεκτρονικά. Αλλά ε, έχω περισσότερη ε, επαφή με ευρωβουλευτές μέσα στο Global Action παρά με συναδέλφους από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μνημειώδης η αλλαγή παρά την ψηφιακή εποχή. Υπάρχει μια μνημειώδης αλλαγή σε ό,τι αφορά τα επιτεύγματα της παγκοσμιοποίησης ε, στο περιβάλλον. Εκεί είναι αναμφισβήτητο ότι η παγκοσμιοποίηση επιτάχυνε πολύ περισσότερο τις εξελίξεις ε, από ό,τι περιμέναμε στον 20ο αιώνα. Τώρα έχουμε μπει στον 21ο αιώνα και οι εξελίξεις είναι πραγματικά ραγδαίες. Αλλά δυστυχώς δεν ε, προοδεύσαμε με αντίστοιχη ταχύτητα στην αντιμετώπιση των ε, οικονομικών προβλημάτων και τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εκεί η απορρίθμιση έλαβε χώρα με εκθετικό τρόπο. Και βέβαια η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία έχει φτάσει σε μια κατάσταση γκροτέσκα πραγματικά, απίστευτη και σίγουρα η Ευρώπη ήταν πολύ χαλαρή ε, στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων ε, της Καρεβικής και της Ανατολής και συμφώνησαν οι υπουργοί μα ε, να ληφθούν κάποια μέτρα, αλλά δυστυχώ η έμπρακτη εφαρμογή του καθυστερεί. Η παγκόσμια εγκληματικότητα χρησιμοποιεί την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κροατία και άλλες χώρες για να ανακτήσει τις ε, δραστηριότητες του λαθρεμπορίου, ε, όπλων, ναρκωτικών, σωματεμπορία και εντείνουν τη διαφθορά στα κράτη-μέλη αυτή οι εγκληματίες του οργανωμένου εγκλήματος. Και παρόλο που γνωρίζουμε την κατάσταση πολύ καλά, οι δράσεις μας είναι πολύ χαλαρές, είναι ελάχιστες και οι πολίτες δεν είναι ανόητοι. Βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των λόγων και των έργων και υπάρχουν μεγάλες ασυνέπειες μεταξύ της ε, θεωρίας και της πράξης. Ο κύριος Τζόνσον μας μίλησε για το πλαίσιο και μας ρώτησε βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο. Ναι, βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο, αλλά μερικοί ταξιδεύουν πρώτη θέση, άλλοι δεύτερη, άλλοι οικονομικοί. Μερικοί έχουν ε, μείνει στην ξηρά και κυρίως αυτοί που έχουν μείνει στην ξηρά, που έχουν χάσει το πλοίο, είναι αυτοί κυρίως από τις χώρες του Νότου. Υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν στην πείνα, στη φτώχεια και στην περιθωριοποίηση. Έμειναν εκτός του πλοίου μας λοιπόν. Ποια είναι λοιπόν η παγκοσμιοποίηση η παγκοσμιοποίηση είναι αυτό που ε, μας δείχνει σε real time τις πληροφορίες από τη Συρία, από την ε, Βόρεια Κορέα. Το Facebook μας δίνει πληροφορίες για το τι συμβαίνει καθημερινά και ταυτόχρονα μας δίνει δυνατότητα ε, για πολύ καλύτερη επαφή και συνεργασία, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις ανησυχίες και τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Γιατί ξέρουμε ότι εκατομμύρια πολίτες δεν γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα, το, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και μάλιστα η συνθήκη της Λισαβόνας ε, στη βασική του δομή είναι δυσανάγνωστο κείμενο περίπλοκο και Είμαι σίγουρη ότι και πολλοί ευρωβουλευτέ αγνοούν το πραγματικό περιεχόμενο τη συνθήκη Λισαβόνα. Πώ να το περιμένουμε λοιπόν τέτοια γνώση από του Ευρωπαίου πολίτε. Οπότε οι πολίτε ε, δεν θα μα κρίνουν από τη ρητορική, από τη νομική ορολογία, αλλά από τα έργα μα, από τα κονδύλια, από τη δράση, από τη φωνή, από την παρουσία. Ανέκαθεν αυτά ήταν τα κριτήρια για του πολίτε. Τα έργα είναι τα πιο σημαντικά. Έχουμε όμως έργα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι. Το θέμα δεν είναι η συζήτηση, το θέμα δεν είναι να εξετάζουμε το παρελθόν. Έχει σταματήσει ο πόλεμος, ευτυχώς έχει σταματήσει αυτή η αιματοχυσία στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται η διέρεση, ο διχασμός, γιατί έχουμε φτώχεια, έχουμε ε, αρρώστιες, ανισότητα και το χειρότερο έχουμε τη δικτατορία των χρηματοπιστωτικών αγορών και των ε, πολυεθνικών. Έχουμε εδώ ένα άρθρο του Guardian που έχει πολύ ενδιαφέρον τίτλο, Θα το διαβάσω στα αγγλικά. Φαίνεται ότι πέρασε ο χρόνος για τη φοροαποφυγή, ότι σταμάτησε πια η δυνατότητα φοροαποφυγής τα 4,2 δισεκατομμύρια τζίρος του Amazon στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, φαίνεται ότι περνάνε από το Λουξεμβούργο και ουσιαστικά δεν φορολογούνται στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα κέρδη από όλες τις πωλήσει. Όταν λοιπόν συζητούμε με τους Αμερικανούς αν η Starbucks, η Google ή η Amazon ή άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να υποφελούνται από την, αυτό το φορολογικό παράδεισο, ενώ οι δικοί μας συμπολίτε επιβαρύνονται φορολογικά εξαιτία των προγραμμάτων λιτότητας και διάσωσης στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίασης, πραγματικά αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούν να δεχθούν οι πολίτες μας να το βουλώνουμε και να μην στυλιτεύουμε τέτοια πραγματικότητα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Γιατί όσο δεν την καταπολεμούμε θα μας υποτιμούν φυσικά οι πολίτες μας όσο και αν συζητούμε για τη σημασία των κοινοβουλίων την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος παίκτη. Θα μπορούσε να είναι παγκόσμιος παίκτη είτε λόγω δράσης είτε λόγω παράληψης. Και δυστυχώς μερικές φορές είμαστε παγκόσμιος παίκτη λόγω παράληψης. Για παράδειγμα, έχουμε μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορά μας ή στα σύνορα με την Τουρκία ή από τη Βόρεια Αφρική. Ποια ήταν η αντίδρασή μας? Σταυρώσαμε τα χέρια και περιμέναμε 8 μήνες το Σεπτέμβριο ε, τη νέα Επιτροπή, το νέο Επίτροπο και τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μεταξύ όμως πώς αντιμετωπίζονται στην ΣΕΟΤΑ οι μετανάστες από μια κυβέρνηση της δεξιάς, αντιμετωπίζονται με λαστιχένιες σφαίρες. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε ε, τόσο ανηλαείς και ταυτόχρονα να ακούμε τον Πάπα Φραγκίσκο που λέ, θα, μας λέει ότι θα πρέπει να είμαστε ανθρωπιστές ενώ φλούμε στα θύματα της φτώχειας και της πείνας. Είναι πραγματικά επονίδιστο να μην λέει κατά τέτοια ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ο Πάπας Φραγκίσκος που είναι πνευματικός ηγέτης να κάνει τέτοιες στοιχειώδει εκκλήσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για στοιχειώδει ελευθερίε και στοιχειώδη δικαιώματα, όπω είναι η ελεύθερη διακίνηση. Αλλιώ ήμασταν πολύ καλά και που ήμασταν και αυτοκυβερνούμασταν πολύ καλά, δεν χρειαζόμασταν Ευρώπη. Γιατί ε, εκχωρούμε την κυριαρχία μας, αλλά θέλουμε ένα αντάλλαγμα. Θέλουμε μια ελεύθερη, ισότιμη, δίκαιη Ευρώπη και πραγματικά μια Ευρώπη αλληλεγγύης και αδελφότητας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, <clears throat> σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία σας. Επόμενος ομιλητής από τη Λιθουανία, κ. Μπάλτσις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ που ε, μας φέρατε. Όσο πιο σφαιρικά γίνονται τα πράγματα, τόσο πιο μεγάλη είναι ανάγκη για συντονισμένη αντίδραση. Η διαπίστωση αυτή πολλές φορές ε, πραγματοποιείται με εντελώς χαοτικό τρόπο ιδιαίτερα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις όπως η χρηματοπιστωτική. Μπορεί όμως να έρθει και με οργανωμένο τρόπο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ την μεγάλη σημασία της ενίσχυσης του ρόλου των κοινοβουλίων των κρατών μελών μέσω συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει το σωστό παράδειγμα που πρέπει να μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο και αναφέρομαι στην ΚΟΖΑΚ, μια από τις πιο επιτυχείς μορφές κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Είχαμε ε, τη συνεργασία αυτή, τη συνάντηση στο Βίλνιους πριν λίγο καιρό και καλό θα είναι να θυμηθούμε λίγο τη συζήτηση ε, στην συνάντηση μετά από 50 χρόνια εν πάση περιπτώσει λειτουργίας της ΚΟΖΑΚ Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής διάστασης. Μην ξεχνάμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία μας δίδει τα σωστά μέσα για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Απαιτείται επίσης ε, σωστή ε, των μέσων που παρέχονται στα κοινοβούλια των κρατών μελών μέσω του διαλόγου. Ο διάλογος ανάμεσα στα κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα υπάρχοντα διακοινοβουλευτικά φόρα έτσι ώστε να πετύχουμε περισσότερους στόχους και αναφέρομαι εδώ σαν παράδειγμα στην ε, Κοζάκ των γυναικών που δημιουργήθηκε στο Βίλνιος που δείχνει ότι μπορεί κανείς να είναι ευέλικτο, σύγχρονος χρησιμοποιώντας ε, τις υπάρχουσες δομές. Και νομίζω ότι το Women's Parliamentary Forum θα μπορέσει στο μέλλον να αποδείξει την αξία του. Πρέπει επίσης να ξεπεράσουμε και τα όρια της Ευρώπης μέσω μιας καλύτερης παγκόσμιας διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. <clears throat> και έχω μια ιδέα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μια πρόταση να κάνω. Την πιθανή δημιουργία μιας κοινοβουλευτική συνέλευσης ανατολικής γειτονίας από χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης όπου αυτό είναι εφικτό βέβαια γιατί υπάρχει μια ειδική πολιτική κατάσταση σε κάποιες από αυτές τις χώρες και των κοινοβουλίων των κρατών μελών φυσικά και του Ευρωπαϊκού Φυσικά Κοινοβουλίου. Μετά από τη συνάντηση κορυφής του Βίλνιους μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η δημιουργία αυτού του κοινοβουλευτικού φόρουμ μπορεί να είναι λειτουργική. Ίσως να είναι υπερβολικά θαραλέο κάτι τέτοιο στην αρχή τουλάχιστον, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε στην αναζωογόνηση ε, κάποιων μικρότερων φόρουμ όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Λιθουανίας, Λετωνίας και Πολωνίας. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει γενικά τις διεθνείς διαστάσεις της κοινοβουλευτικής συνεργασίας. Αυτό απαιτείται και σε παγκόσμιο επίπεδο να αναπτυχθούμε αλλά να δράσουμε τοπικά. Και ένα τρίτο θέμα είναι η ανάγκη ενίσχυσης των διακοινοβουλευτικών οργανώσεων επί τη βάση κοινών στόχων και συμφερόντων. Και εδώ έχουμε τα Globe International και τα Globe Europe και είμαι και αντιπρόεδρος αυτών των δύο δομών. Σαν παράδειγμα θέματα αναθεώρησης των νομοθεσιών γύρω από το περιβάλλον σε 66 χώρες να λοιπόν πώς μπορούν ε, οι βουλευτές από διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές ιδεολογίες να πετύχουν κοινού στόχους στον τομέα του περιβάλλοντος. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες ε, συνεργασίας, όχι με βάση ε, την πολιτική προέλευση αλλά τα συμφέροντα των χωρών ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης με ειρηνικό και αποτελεσματικό τρόπο. Πολύ ωραία. Τελευταίοι δύο μιλητές. Ο κύριος Καμέλο Αμπέλα και ο κύριος Ζάρο. Ο κύριος Καμέλο Αμπέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση και επίσης θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Γιώχανσον για την ομιλία του. Πιστεύω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση μπορεί να μας βοηθήσει για να ε, παρουσιάσουμε το πώς ακριβώς ε, εργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα. Στο εθνικό επίπεδο σε επίπεδο κυβέρνησης και επίση και σε ε, διεθνή φόρα. Εξάλλου, μπορούμε να κάνουμε και την εξής ερώτηση. Τελικά, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις. Τις λαμβάνουν οι κυβερνήσεις, μήπω τα εθνικά κοινοβούλια, οι διεθνείς οργανισμοί. ή μήπω οι αποφάσεις λαμβάνονται από άλλες ε, δυνάμεις. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν για να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η συνεργασία όπως και οι προσπάθειες όλων αυτών των δυνάμεων. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι ότι πράγματι είναι αλήθεια ότι ζούμε σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ότι η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει όλες τις χώρες, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι οι εσωτερικές εθνικές αποφάσεις επηρεάζουν, ασκούν επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα, αυτό που είπε ο κύριος Κόβαξ, όπου αναφέρθηκε στην Αραβική Άνοιξη. Σε πολλές περιπτώσεις η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε από την ιδιωτική πρωτοβουλία όπου οι άνθρωποι ε, στράφηκαν κατά του ε, κατεστημένου μιας ε, χώρας. Αυτοί ξεκίνησαν όλες αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι οι εθνικές αποφάσεις ασκούν παγκόσμια επιρροή. Και τέλος πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ασκούμε πολιτική προς όφελος των πολιτών. Η δουλειά μας είναι να κατανοήσουν οι πολίτες τη σημασία της δουλειά μας, να κατανοήσουν ότι υπηρετούμε αυτούς. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Εμείς ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ως στόχο να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε τη φτώχεια. Έχουμε όμως και άλλους στόχους. Μερικές φορές πιστεύω ότι αυτοί οι δύο παράγοντες ε, αντιπαλεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολλές φορές για να εξαλείψει κανείς τη φτώχεια φτώχεια πρέπει να ε, προβλέψει εθνικά επιδόματα που όμως με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες. Και εδώ υπάρχει ακριβώς αυτή η αντίφαση. Αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες, ε, πρέπει όμως να εξαλειφθεί η φτώχεια. Βλέπουμε πολλές φορές ότι οι αποφάσεις ε, που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο οδηγούν ακριβώς σε τέτοιου είδους αντιφάσεις και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την εσωτερική συζήτηση για το πώς ακριβώς τα κράτη-μέλη αλλά και οι κυβερνήσεις μπορούν να συνεργαστούν, αναφέρομαι στις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, που πρέπει να λειτουργούν παράλληλα γιατί κανένα από τα δύο δεν μπορεί να υποκαταστήσει το άλλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε κοινό μέτωπο. Ο κύριος Γιώχανσεν έθεσε μια πολύ σημαντική ερώτηση σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε πολυμερή φόρα ή όχι. Εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία. Ε, πολλές φορές πάμε σε αυτές τις ε, διεθνείς ε, συναντήσεις όπου αυτά τα πολυμερή φόρουμ, η φόρα ε, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Έχουμε την Διεθνή Κοινοβουλευτική Ένωση, πολλές άλλες ε, συνελεύσεις. Αλλά τελικά αυτό που γίνεται σε αυτές τις συνελεύσεις δεν ακούγεται πολύ δυνατά. Δεν ακούγεται σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για να παραμείνουμε σημαντική να έχουμε περισσότερη συνεργασία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση αυτής της συνάντησης και για τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης με τον οποίο έχουμε μοιραστεί πολλά τα τελευταία χρόνια. Άκουσα τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων και νομίζω ότι τέσσερα είναι τα βασικά θέματα τα οποία είναι τα κομβικά αν θέλετε που πρέπει να προκαλέσουν την προσοχή μας. Πρώτον, θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι γίνεται με τον μεγάλο αριθμό των διακοινοβουλευτικών διεθνών οργανώσεων, τον συντονισμό των εργασιών αυτών και θα πρέπει οι εργασίες τους να εκτιμηθούν σωστά από τους πολίτες. Δεύτερον, θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις στην έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στα διεθνή κοινοβουλευτικά όργανα και τα κοινοβούλια των κρατών μελών δεν υπάρχει σωστό συντονισμός και αυτό δημιουργεί συγκεκριμένες δυσλειτουργίες. Τρίτον, θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις ε, για την έλλειψη ε, μερικές φορές ε, εμπιστοσύνης των κοινοβουλίων των κρατών μελών προς τις διεθνείς κοινοβουλευτικές οργανώσεις. Πρέπει να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και τέλος είναι απαραίτητο να υπάρξει μια προσπάθεια παιδαγωγική σε εισαγωγικά γνωστοποίησης, μια πολιτική γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων των οργανώσεών μας έτσι ώστε να γνωρίζουν καλύτερα οι πολίτες τα θέματα της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας που οδηγούν στην βελτίωση της δημοκρατίας. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές ε, δραστηριότητες τις οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και για τις παρεμβάσεις τους και κυρίως τον κύριο Τζόνσον. Εγώ δεν θέλω να περάσω σε μια ιδιαίτερη πολεμική σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πω εδώ ότι η Guardia Civil έχουν προσπαθήσει και έχουν διασώσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος διώκεται και έχει υποστεί ε, πάρα πολύ, ε, ε, πάρα πολύ κόσμο. Θυμίζω ότι δεν είναι μόνο η ισπανική η Θέουτα και η Μελίγια, αλλά είναι το νότιο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τζόνσον έχει το λόγο. Δεν φαντάζομαι να περιμένετε τώρα να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, με ξεπερνάει κάτι τέτοιο. Πάντως, πολλοί από εσά στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης επανήλθατε στις ευθύνες, στην ευθύνη των Εθνικών Κοινοβουλίων και νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη εποπτεία και να συμβάλλουν πιο πολύ με προτάσεις ε, στις ε, διαπραγματεύσεις στις διεθνείς οργανισμούς. Χθες ε, ήμουν στο Βουκουρέστι και συζήτησα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και με τον πρόεδρο της Βουλής. Και συζητήσαμε πώς στη Ρουμανία η Εθνική Βουλή προσπαθεί να επηρεάσει και να έχει λόγο και στις διεθνείς σχέσεις. Και για 7 ολόκληρα χρόνια είχαμε ε, διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής και έχουμε πια και νομοθεσία στη Ρουμανία με συμφωνία της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας που καθιστά υποχρεωτικό για την κυβέρνηση να ε, διαβουλεύεται σε για πολλούς τομείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ξεκινήσει οι διεθνείς διαπραγματεύσεις ε, σε διεθνές επίπεδο. Και θα πρέπει το Κοινοβούλιο, το Ρωμανικό Κοινοβούλιο να δώσει διαπραγματευτική εντολή στην κυβέρνηση. Αυτό πια είναι υποχρεωτικό και είναι και πολύ καλό παράδειγμα το πώς ε, μπορούν τα κοινοβούλια να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων, έχουν λόγο από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Γιατί έτσι πραγματικά θα επηρεάσουν και όλη τη διαπραγματευτική διαδικασία και τη θέση της κυβέρνησης. Και θα μπορούσαν πολλές άλλες χώρες, αν δεν έχουν παρόμοιο μοντέλο, να μιμηθούν το παράδειγμα της Ρουμανίας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι και δεν το είπα ρητά στην παρουσίασή αλλά ήταν ε, έμεσα κάτι που υπήρχε, ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός των ε, διακοινοβουλευτικών οργανώσεων και είναι αναπόφευκτη η επικάλυψη μερικέ φορέ, αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει κάτι είναι δύσκολο να σταματήσει. Και έγιναν κάποιε απόπειρε ε, να κλείσουν μερικές διακοινοβουλευτικέ οργανώσει και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ξέρετε όταν ε, έχετε την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση, βλέπετε τι δύσκολο ήταν να ε, διεκπαιρεωθεί αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχουμε δύο διδάγματα εδώ να αντιλήσουμε. Θα πρέπει να το σκεφτούμε δύο φορές πριν αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο. Να εξασφαλίσουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Και επίσης, όπως είπε ο συνάδελφος, θα πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και οργανώσεων. Εμείς ε, σε επίπεδο διακοινοβουλευτικής ένωσης ε, εφαρμόζουμε αυτό το μήνυμα και τα τελευταία δύο χρόνια στις συνελεύσεις μας δίνουμε το λόγο και σε εκπροσώπους αυτών των οργανώσεων. Τους έχουμε προσκαλέσει και συζητούμε μαζί τους τα θέματα, κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε τουλάχιστον ενημερώνονται και αυτές οι οργανώσεις για το έργο της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Έτσι βελτιώνεται ο συντονισμός και πιστεύω ότι αυτή θα είναι η απαρχή μεγαλύτερης συνέργειας και περιορισμού των επικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων. Επίσης, να επανέλθω σε κάτι που αναφέρατε πολύ, το θέμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ε, που είναι πολύ πιο ισχυροί από τις ίδιες κυβερνήσεις. Διεθνή συνεργασία, το τραπεζικό σύστημα για παράδειγμα. Και εμείς το διαπιστώσαμε αυτό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όταν η Διακοινοβουλευτική Ένωση πηγαίνει στα Ηνωμένα Έθνη και διαπραγματεύεται προσπαθώντας να καθορίσει το ρόλο των κοινοβουλίων στα Ηνωμένα Έθνη, αυτό είναι πολύ απλό, το έργο είναι πολύ απλό σχετικά όταν, ε, σε σχέση με με, τα, τις, ε, με τον Woods, τα Ιδρύματα του Bretton Woods ή με, την, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πολύ πρόσφατα καταφέραμε να ε, μπούμε στην, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στο, στην Παγκόσμια Τράπεζα όμως και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν ε, έχουμε... δεν έχουμε εξασφαλίσει το παρόν. Παρόλο που υπάρχει κοινοβουλευτικό δίκτυο, είναι όμως κοινοβουλευτικό δίκτυο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Δεν είναι ανεξάρτητη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που θα καθιστά υπόλογη την Παγκόσμια Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν ε, σημαντική διαφορά. Και κάτι άλλο, την τελευταία διετία η Διακοινοβουλευτική Ένωση έκανε μία μελέτη για το ρόλο που έχουν τα κοινοβούλια σε σχέση με τα δάνεια και τις πιστώσεις που δίνει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει κάποια διαδικασία που να εξασφαλίζει κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών των διαδικασιών. Και θα πρέπει αυτά τα δάνεια και πιστώσεις να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο, όπως γίνεται με τον προϋπολογισμό. Η μελέτη λοιπόν που καταρτήσαμε από κοινού με το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατέληξε στο πόρισμα ότι σε μεγάλο βαθμό τα κοινοβούλια δεν αναμειγνύονται σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε η μελέτη που εμείς την ε, συγγράψαμε έκανε μια σύσταση με βάση τις βέλτιστες πρακτικές κάποιων χωρών θα πρέπει να υπάρχει και ανάμειξη και συμμετοχή των κοινοβουλίων. Τότε το, δημοσιο... το Μισματικό Ταμείο ε, εγκατέλειψε τη μελέτη, αφαίρεσε τη συμμετοχή του και βλέπετε ότι δεν αναφέρεται πουθενά στους ε, ε, συντάκτες. Και η Παγκόσμια Τράπεζα με πολλή απροθυμία συνέχισε τις εργασίες. Βλέπετε πόσο απρόθυμα είναι τέτοια θεσμικά όργανα απέναντι στην κοινοβουλευτική συμμετοχή στις διαδικασίες τους. Πάντως, ε, παραλαμβάνω, εσείς ε, μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα διαβήματα προς τους ε, θεσμούς αυτούς. Και με εξέπληξε πριν από πολλά χρόνια, όπου όταν ανακάλυψα ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση μέχρι το 2000 δεν είχε κάνει καμία συζήτηση, ούτε σε Επιτροπή, ούτε στην Ολομέλεια, για την συμβολή, τη συνεισφορά της Γαλλίας στην Παγκόσμια Τράπεζα. Παρόλο που η Γαλλία είναι σημαντικό συνεισφορέα στην Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ουδέποτε δεν είχε ελέγξει την γαλλική αυτή συνεισφορά στην Παγκόσμια Τράπεζα και δεν είχε εξετάσει καν την πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κατάσταση άλλαξε το 2000, αλλά μέχρι το 2000 δεν είχε γίνει τίποτα. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι εναπόκειται στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, κάνουν, να εξασφαλίσουν πολύ πιο συστηματική και ενεργό συμμετοχή βελτιώνοντας τη σημερινή κατάσταση. Αυτή είναι η σύσταση. Περισσότερη συμμετοχή, περισσότερο έργο. Και μια και σήμερα εκπροσωπώ εδώ τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, την IPU, θα ήθελα να επαναλάβω ότι όλα αυτά τα χρόνια χάρηκα ιδιαίτερα την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχει και τεράστιο δυναμικό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο, δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Υπάρχει χώρος για πολύ περισσότερη συνεργασία. Και από πολιτική άποψη και η δική μας Διακοινοβουλευτική Ένωση χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα έλεγα μάλιστα ότι Πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κερδίσει από στενότερη συνεργασία με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και ελπίζω να μην το κρίνετε αλαζονικό. Το κάνουμε ούτως ή άλλως για εμπορικά ζητήματα. Γιατί όμως θα σταματήσουμε εκεί. Μπορούμε να έχουμε ακόμη πιο στενή συνεργασία και για πολλά άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Ε, Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω πώς ε, αισθάνεστε εσείς, αλλά η δική μου εντύπωση είναι ότι είχαμε μια ιδιαίτερα ενημερωτική συνάντηση, πολύ ενδιαφέρουσα για όλους, μας ενέπνευσε όλους η συζήτηση σήμερα το πρωί και πρέπει να πω ότι από την πρώτη παρέμβαση μέχρι και την τελευταία ακούσαμε Με συγχωρείτε, διακόπτει ο πρόεδρος. Έχετε την καλοσύνη να κλείσετε εσείς παρακαλώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, από τη μία πλευρά ακούσαμε αναλύσεις που ενέπνευσαν πάρα που τους ε, προκάλεσαν έτσι πολλές καινούργιες σκέψεις. Από την άλλη όμως ακούσαμε και προτάσεις και έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι μάλιστα από εσάς ε, καταγράψατε αυτές τις ε, προτάσεις. Ό,τι λοιπόν συζητήθηκε σήμερα το πρωί νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό πρελούδιο για σήμερα το απόγευμα όπου θα ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με τα θέματα που εθίγησαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και θέλω να πω και κάτι. ορισμένα από αυτά που συζητήσαμε σήμερα, ορισμένα εξ αυτών εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο σε εθνική δικαιοδοσία. Άρα δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε με τα του οίκου μας. Κάποιος ε, συνάδελφος ε, από τη Λετωνία διαμαρτυρήθηκε για το ότι η απόφαση ένταξης της χώρας στο ευρώ ελήφθη μόνο από την κυβέρνηση και κανέναν άλλον. Κοιτάξτε όμως, ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις ε, εθνικές ε, διαδικασίες λήψη αποφάσεων, ε, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη συμμετοχή της χώρας σε μια ευρωπαϊκή απόφαση ή όχι. Όπως γνωρίζετε, οι εθνικοί μηχανισμοί λήψη αποφάσεων προβλέπονται στο σύνταγμα της κάθε χώρας και δεν μπορούν να επικοτισταθούν οι μηχανισμοί αυτοί από άλλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι άλλο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαμαρτυρόμεθα για την επικυριαρχία του ε, Συμβουλίου Υπουργών, ε, διαμαρτυρόμεθα για την αποδυνάμωση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως για τον έλεγχο και το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στα κράτη-μέλη, γι' αυτό το θέμα αρμόδια είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι εκείνα που φέρουν την ευθύνη άσκησης ελέγχου στη κυβέρνησή τους είναι εκείνα που καλούνται να αποφανθούν κατά πόσο είναι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι με βάση το κοινοτικό δίκαιο ή οτιδήποτε άλλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι σύνομοθέτης και ελέγχει μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δικαιούται να ελέγχει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ορισμένοι ε, τοποθετήθηκαν για το θέμα των ε, μηχανισμών, των φορολογικών μηχανισμών. Και έχετε δίκιο, τα φορολογικά εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσες δυσκολίες υπάρχουν ε, στην Ευρώπη στο να καθορίσουμε ένα κοινό φορολογικό πλαίσιο ή αν θέλετε στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους φορολογικούς παραδείσους ανά τον κόσμο. Είναι σαφές ότι τα φορολογικά θέματα ε, θα πρέπει, αν το επιθυμήσουν τα κράτη-μέλη, να εξευρωπαϊστούν μετά από αποφάσεις αυτών των κρατών μελών. Εγώ λοιπόν θεωρώ και λέω, ισχυρίζομαι, ότι ότι οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες στα κοινοβούλια και όχι το αντίθετο. Κατόπιν τούτου πρέπει να σας πω, νομίζω η Πορτογαλία το είπε αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κρίσης δεν απέφυγε λάθη δεν υπέπεσε σε λάθη όσον αφορά στο μνημόνιο, στα μνημόνια που υπογράφησαν. Μα πώς να υποπέσουμε σε λάθος αφού δεν συμμετείχαμε. Ήμασταν εκτός της όλης διαδικασίας. Κατά την αντιμετώπιση της ε, κρίσης, δυστυχώς υπήρχαν ελάχιστοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Και αυτοί που υπήρχαν, όσοι υπήρχαν, ήταν και σε δύο επίπεδα. Και αν θέλετε, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Προκλήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί από τότε που εισήχθη το ευρώ ως κοινό νόμισμα, οτιδήποτε έχει σχέση με κοινό νόμισμα από τότε δηλαδή που ελήφθηκε η απόφαση στη συνθήκη του Μάστριχτ, δυστυχώς έκτοτε δεν υπήρξε καμία άλλη συλλογική ανάληψη αυτινών. Στη συνθήκη του Μάστριχτ αναφέρεται ότι μέχρι την τρίτη φάση της νομισματικής ένωσης οι αρχές της πολιτικής ένωσης πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτό λέει η συνθήκη του Μάστριχτ. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να συντονίσουμε εκείνα τα πολιτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για ε, να αποφύγουμε την οικονομική κρίση. Συντονίζουμε δηλαδή μόνο τα πολιτικά εργαλεία για να αποφύγουμε μια ε, διάδοση, περαιτέρω διάδοση της, της κρίσης. Διαμαρτυρόμεθα για την πρωτοκαθοδρία των αγορών, αλλά μόνο ε, επειδή ακριβώς προέκυψε η κρίση, μόνο για αυτόν τον λόγο τελικά καταλήξαμε στην τραπεζική εποπτεία. Το 2010, θα ξέρετε, η πρόταση τραπεζικής εποπτείας απέτυχε, απορρίφθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών. Το 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησαν τον έλεγχο στατιστικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Όμως η Υπουργή Οικονομικών, το ΕΚΟΦΗΝ, διαφώνησε. Το 2010, μόλις το 2010, εκφράστηκε η πολιτική βούληση να ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο τα στατιστικά δεδομένα που αποστέλουν τα κράτη-μέλη. Και τώρα συζητάμε για την Τραπεζική Ένωση ως απάντηση στην κρίση, παρότι η Τραπεζική Ένωση πριν από 20 χρόνια τουλάχιστον αντιμετωπίζεται ως λογική συνέπεια της Νομισματικής Ένωσης. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω το εξής, ότι παρακαλώ η πολιτική βούληση και η προθυμία για ανάληψη πολιτικών δράσεων, αυτή η βούληση να προβάλλεται προς τα έξω, να προβάλλεται στην κοινή γνώμη και απέναντι στις κυβερνήσεις. Αυτό όμως να γίνεται έγκαιρα, όταν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, όχι εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε αλλιώς χάνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, χάνουμε την αξιοπιστία μας για την πολιτική μας πράξη. Και κάποιος εξημών ε, είπε κάτι που θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω, ε, είπε λοιπόν ότι επιθυμούμε την κοινοβουλευτική διάσταση να παρισφρήσει αυτή στην παγκοσμιοποίηση χωρίς όμως παράλληλα να περικοπούν τα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων. Επαναλαμβάνω, λέει ο πρόεδρος, κοινοβουλευτική διάσταση στην παγκοσμιοποίηση χωρίς περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Ε, και διερωτώ με, πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μερικές φορές δεν θίγονται καν θέματα χρηματοπιστωτικών αγαρών, χρήματος, τεχνολογίας. Εάν ο καθένας θέλει την εθνική του κυριαρχία για να διαμαρτύρεται εκ των υστέρων επειδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές, η τεχνολογία και οι αγορές καθορίζουν την ε, πολιτική μας δράση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ε, ο στόχος μας, δεν είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερα να μοιραζόμαστε μία κυριαρχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί να χάσουμε πλήρως την κυριαρχία μας και να είμαστε έρμεα άλλων ή όμοιροι άλλων. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούμε και όχι να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε λύσεις. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις ε, που να μην είμαστε παρόντες. Αλλά ε, δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις όπου ε, τις αποφάσεις τις παίρνει ο μόνος του. Πιστεύω λοιπόν ότι μερικές φορές όταν μιλάμε για την εθνική ευθύνη υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρώπη δεν ευθύνεται. Μερικές φορές όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή ευθύνη στα κράτη μας προκαλούμε την εντύπωση ότι εμείς ε, δεν είχαμε κανένα λόγο. Και Τώρα που γίνεται λόγος για την παγκόσμια διακυβέρνηση, πολύ συχνά και ως πολιτικοί προκαλούμε την εντύπωση ότι άλλοι αποφασίζουν για εμάς και εμείς δεν συμμετέχουμε καθόλου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διαμορφώσουμε συστήματα όπου θα είναι απόλυτα σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί καμία απόφαση χωρίς τη συμμετοχή των κοινοβουλίων. Από αυτή λοιπόν τη συζήτηση εγώ εξάγω δύο συμπεράσματα. Γιατί δεν μπορούμε σε όλες αυτές τις ε, συναντήσεις μας που είναι έτσι παγκόσμιας ε, διάστασης να εκφράζουμε τις απόψεις ε, των κρατών μελών και γιατί όταν γίνονται ε, συζητήσεις παγκόσμιου ελληνικούς. Δεν συζητάμε στα εθνικά μας κοινοβούλια για αυτά που πρόκειται να συναντηθούν σε αυτές τις συναντήσεις και μάλιστα μπορούμε και να συζητάμε με video conferencing, με τέτοιου είδους συζητήσεις. Γιατί δεν απαιτούμε οι κυβερνήσεις στις ε, αντιπροσωπείες ε, να συμπεριλαμβάνουν αναγκαστικά ε, εκπροσώπους των κοινοβουλίων. Ποιος μας εμποδίζει να το απαιτήσουμε αυτό. Ποιος μας εμποδίζει να ζητήσουμε κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί και να πει στον Υπουργό του των Εξωτερικών κοιτάξτε αν στείλετε ας πούμε μία αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ή οπουδήποτε αλλού οπωσδήποτε θα συμπεριλαμβάνονται ε, στην Επιτροπή αυτή και μέλη της δικής μας της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σε τελική ανάλυση ποιος εμποδίζει ε, υπουργό οι ε, κυβερνήσεις ε, να έρχονται στα κοινοβούλια για να συζητήσουν τα θέματα που θα θυγούν σε μια διεθνή συνάντηση και μάλιστα εκ των υστέρων να επανέρχονται στα κοινοβούλια και να τα ενημερώνουν για το τι ακριβώς διαδραματίστηκε. Στη τελική ανάλυση ποιος μας εμποδίζει όπου εμφανιζόμαστε όλοι από κοινού, να ε, συνδεόμαστε με τα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν, ε, χωρίς να είναι απαραίτητο μάλιστα να γίνονται και όλα αυτά τα ταξίδια. Σήμερα λοιπόν εμείς είπαμε εδώ ότι για την ε, συνεδρίαση των G20 θέλουμε η μερίσια διάταξη να μας δίδεται μία εβδομάδα νωρίτερα, να τη συζητάμε αυτή την ημερήσια διάταξη, να αποφασίζουμε για ένα κοινό ψήφισμα και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας που φιλοξενεί τη συνάντηση των G20 θα είναι εκείνος ο οποίος πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση θα ανακοινώνει στους μετέχοντες των G20 αυτό το ψήφισμα. Αν θέλετε αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρώτο βήμα και ξέρετε, αν γίνει, αυτό θα προκαλέσει την κοινή γνώμη. Και αυτό πάλι ευαισθητοποιεί τους πολίτες και προκαλεί και τη συμμετοχή των πολιτών. Πολλές από τις ε, προτάσεις που κάνετε στην Τρόικα, έρχομαι στην Τρόικα ως τελευταίο παρατήρηση. Κοιτάξτε, η Τρόικα είναι διακυβερνητικό όργανο και ήταν απαραίτητο γιατί δεν υπήρχε τίποτα το αντίστοιχο. Το μόνο που είχαμε ήταν η συμμετοχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν λοιπόν αφήναμε να βοηθήσει μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό πρώτον θα είχε χορηγήσει μικρότερα κονδύλια με ε, μεγαλύτερα, υψηλότερα επιτόκια σε συντομότερο χρονικό διάστημα και πιο αυστηρά προγράμματα. Άρα δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να εξευρωπαίσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όμως δεν είχαμε απαραίτητα εργαλεία για κάτι τέτοιο. Και αυτό που λέμε τώρα είναι το εξής όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ελέγχονται και να νομιμοποιούνται από τα κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να παρισφρεί και να εφαρμόζεται στα ε, εκτελούμενα προγράμματα. Αυτά προφανώς μακροπρόθεσμα με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Ίσως ε, κάποια μέτρα που ελήφθησαν να ε, λαμβάνονται παρόλα αυτά. Ίσως. Όμως θα υπήρχε διαφάνεια, συμμετοχή, έλεγχος και τα αποκαλούμενα rules of procedure. Δεν είναι δυνατόν ούτε στη τελική ανάλυση μας ενδιαφέρει να στυλιτεύσουμε τα πάντα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα για το μέλλον. Και τελευταία μου πρόταση Πολλές από τις συνέπειες, ε, πολλά από τα συμπεράσματά μας ως απάντηση στην κρίση ε, δεν μπορούν συμπεράσματα αυτά δικά μας να υλοποιηθούν χωρίς να τροποποιηθούν οι συνθήκες. Και ερωτώ, Θέλετε, τολμάμε να ζητήσουμε αλλαγή των συνθήκων. Γιατί αν το θέλουμε αυτό, ξέρετε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ομοφωνία. Είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε στους πολίτες και να τους πούμε αυτές είναι οι προτάσεις μας ως κοινοβούλια για την ενίσχυση των κοινοβουλίων, την ενίσχυση της διαφάνειας, την ενίσχυση του ε, δημοκρατικού ελέγχου της ε, δυνατότητας ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουμε και κοινωνόμισμα. Το τολμάμε αυτό ή από την άλλη μόνοι μας το μόνο που κάνουμε είναι να υπεραμεινόμενθα της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί αν δεν εξεγερθούμε και δεν πάμε στους πολίτες και δεν θελήσουμε να τους συμπεριλάβουμε, ποτέ δεν θα έχουμε τη δημοκρατική πλειοψηφία για να επιτύχουμε αυτά που όλοι μας κρίνουμε απαραίτητα. Γι' αυτό αυτή η συνάντηση σήμερα είναι καθοριστική σημασίας. Δεν πρόκειται απλά για αρμοδιότητες. Αν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως κοινοβούλιο, δεν θα έχουμε διαφάνεια και οι κυβερνήσει θα αποκτήσουν περισσότερες εξουσίες για τη τελική ανάλυση κάποιο καλείται να κάνει κάτι. Αν δεν κάνουμε κάτι εμεί, θα κάνουν οι άλλοι. Και απλά με τον τρόπο αυτό σε επίπεδο κυβερνητική συνεργασία, θα ε, συστήνονται μία επιτροπή μετά την άλλη οι οποίε επιτροπές αυτέ, απλά θα αποδυναμώνουν και το κοινοβούλιο και του πολίτε. θα αγνοούν του πολίτε. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα θέματα που εθίγησαν εδώ πραγματικά ήταν εντυπωσιακά και προτείνω να μην ε, σταματήσουμε σήμερα αυτή η συνάντησή μας, να μην σταματήσει εδώ, να συμπεριλάβουμε πάρα πολλά θέματα που θα συζητάμε, το διαδίκτυο, την κοινοβουλευτική δημοκρατία και άλλα, γιατί όπως ακούσαμε υπάρχει ένα μοντέλο ε, του κοινοβουλευτισμού και της κοινοβουλευτικής διάστασης και σε σχέση με τον ΠΟ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η IPU μπορεί να ε, υιοθετήσει αυτό το μοντέλο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης που υπάρχει ε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μπορεί να το μιμηθεί αυτό το μοντέλο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε και τα, σήμερα το απόγευμα σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί θεωρώ ότι η συζήτησή μας ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και ο κάθε ένας από εσάς κατέθεσε νέες προτάσεις. Και τώρα καλή σας όρεξη. Yes. We are going for, we are going for lunch together. Uh, please follow us. It's downstairs on the zero floor.